Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne... συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, άρχεται η συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας. Έχετε την ημερήσια διάταξη. Μπορεί να εγκριθεί αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, ενστάσεις. Δεν υπάρχουν. Εγκρίνεται. Ανακοινώσεις Προέδρου δεν υπάρχουν. Περνάμε στο σημείο 3 προπαρασκευή για την αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 μετά από τις ευρωεκλογές. Τοποθέτηση του Ευρωκοινοβουλίου στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εισηγητής ο κύριος Μαρινέσκου έχει τον λόγο. Παρακαλώ. Eh, Πρόεδρε. Eh, αφού Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρουσιάστηκαν, υπευλήθησαν ε, τροπολογίες για την έκθεση αυτή και έχουμε ήδη συζητήσει και προετοιμάσει κάποιες ε, συμβαστικές με τις πολιτικές ομάδες. Ε, δεν φαντάζομαι ότι θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, τουλάχιστον προς το παρόν. και συζητήσαμε επίση σχετικά με την ανάκτηση κονδυλίων τα οποία είχαν μεταφερθεί προς την εύση. Σχετικά κυρίως ε, με την επανεξέταση του προϋπολογισμού όπου είχαν, ε, είχαν ζητηθεί συμπληρωματικά κονδύλια για την Connecting Europe Facility. Επίση είχαν υποβληθεί στοιχεία σχετικά με τους διαγωνισμούς που μόλις είχαν ολοκληρωθεί. Είναι επίσης σημαντικό να έχουμε πορούς για το Γαλιλαίο. Ε, διαστημικό, πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, πάρα πολύ σημαντικό για τις ε, υπηρεσίες μεταφορών μας. Πρέπει να επιχειρήσουμε επίσης ένα συντονισμό για την περιφέρεια του Δούναβη αλλά και της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας δημιουργώντας ενέργειες μεταξύ των ε, μακροπεριφερειών αυτών. Και στο πλαίσιο της αναθεώρησης ε, προσπαθούμε για το μέλλον να έχουμε διαβιβάσεις, μεταβιβάσεις για τα πλεονάσματα, δηλαδή για κονδύλια που δεν έχουν μεταφερθεί εντός ενός έτους. Ώστε να μπορούμε να εκτελούμε πλήρως τον προϋπολογισμό που ενεκρίθη το 2013. Και ελπίζοντας ε, βεβαίως να φτάσουμε σε μια εκτέλεση του επίπεδου του 100%. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά σημεία που ήθελα να σημίσω. Να θυμίσω, με συγχωρείτε. Υπάρχει και το θέμα βεβαίως του τουρισμού που δεν το ξεχνούμε. Ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους τους εισηγητέ των άλλων πολιτικών ομάδων για τη στήριξη και για την εξαιρετική συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ισκιώδης εισηγητέ πρώτα. Πυρίνσκι παρακαλώ. Δεν παρίσταται. Ο κύριος Τομάσικ παρακαλώ. Ούτε και αυτός παρίσταται. Ντομινίκλη και παρακαλώ. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αφού δεν έχουν έρθει, τότε θα έχω εγώ περισσότερο χρόνο για να μιλήσω. Ευχαριστώ τον Μαριάν, ήταν εξαιρετική η δουλειά που έκανε και αγαστή συνεργασία και με τους σκιώδεις εισηγητές. 13 συμβαστικές είναι ε, το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας ε, και της υποστήριξής μας. Νομίζω δεν θα υπάρχει καμία δυσκολία. Θα ήθελα να σχολιάσω πρώτα απ' όλα τη δυσκολία συγκρότηση επταετού δημοσιονομικού πλαισίου στην Ευρώπη, όταν βλέπουμε ότι με τα βία μπορούμε να διαχειριστούμε αυτά που θα συμβούν τον επόμενο μήνα. Είναι τόσο ραγδαίε οι εξελίξει που ε, ακόμη και ετησίω είναι καθίσταται δύσκολο να διαχειριστούμε τον προπολογισμό. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο περιοριστικό είναι ένα επταετέ πλαίσιο Ταυτόχρονα οι διαρκείς περικοπές ε, κονδυλίων και η ε, σημερινή κατάσταση δυσχερούν έτσι περαιτέρω το έργο μας. Δεν πρόκειται για μια απλή αναθεώρηση Πρόκειται για ανασυγκρότηση του πλαισίου και ελπίζω να έχουμε πιο αποτελεσματικά, πιο επιχειρησιακά μέτρα από πλευρά ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ε, το βασικό πρόβλημα είναι η ανάπτυξη στην Ευρώπη. Είναι αδύναμη, πρέπει να την υποστηρίξουμε και θέλουμε να προωθήσουμε άμεσα την ανάπτυξη με συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες, υποστήριξη των οικονομικών δραστηριοτήτων ε, των πολιτών και ε, βλέπουμε ότι είναι απαραίτητη η χρηματοδότηση των σχεδίων υποδομής. Όλοι οι Σκιώδης και ο Μαριάν στην παρουσίασή του τόνισαν ότι η κατάσχεση από το από το μηχανισμό συνδέοντα την Ευρώπη, η ΣΕΦ, ε, είναι κάτι που ε, μας απογοήτευσε ιδιαίτερα και είδαμε ότι έγιναν ε, δύο διαφορετικές ε, προσκλήσεις υποβολής ε, προσφορών και σχεδόν εξαντλήθηκαν τα κονδύλια. Βλέπουμε ταυτόχρονα όμως πόσο δυναμικός και πόσο μεγάλο δυναμικό έχει αυτός ο μηχανισμός. Θα έρθει η Επίτροπος Μπούλς και θα μας εξηγήσει σε λίγο ποια είναι τα σχέδια του ΕΕ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών. Θα δούμε αν τα προγράμματα που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή αυτή η δομή που διαχειρίζεται τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων όντω προσφέρουν μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και αν ανταποκρίνονται στι ανησυχίε τη Επιτροπή Μεταφορών του Κοινοβουλίου. Εάν υπάρχει, αν τηρείται δηλαδή η αρχή της προσθετικότητας, δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε δημοσιονομικά εργαλεία εκτός επιδοτήσεων και η αναδιάταξη των κονδυλίων από το ΣΕΦ ε, σίγουρα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα προγράμματα υποδομής της Ευρώπης. Ε, πώς θα αντέξουμε τρία χρόνια ακόμη με άδεια τα ταμεία, ε, μιλώντας φυσικά για τις επιδοτήσεις, για τη χρηματοδότηση και δεδομένου του ότι χρειαζόμαστε μεγάλα προγράμματα υποδομής ε, για την Ευρώπη και δεν θα έχουμε δυστυχώς ε, το, το, τη μόχλευση που χρειαζόμαστε χάρη στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε την Επίτροπο διότι ε, αυτό σχετίζεται άμεσα με την συγκρότηση του δημοσιονομικού πλαισίου και την έκθεση του Μαριάν. Ε, Επίση, έχουμε την επιπρόσθετη αρμοδιότητα στον τομέα του τουρισμού για την Ευρώπη, όμω εκεί δεν έχει σημειωθεί καμία συγκεκριμένη πρόοδο. Κλείνοντα, να σα πω πω κατά πάσα πιθανότητα αυτό το εργαλείο του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου πλέον δεν ανταποκρίνεται στην ουσιαστική διαχείριση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δημοσιονομικό κανονισμό πλέον δεν ανταποκρίνεται στι ανάγκε μα και είμαστε όμοιροι ε, αυτού του συστήματο ε, που δυστυχώς θυμίζει το πενταετές ε, σοβιετικό πλαίσιο ε, που σίγουρα όλοι γνωρίζαμε ότι ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί και χρειαζόμαστε λοιπόν αναθεώρηση, πραγματική, ουσιαστική ανασυγκρότηση του πλαισίου ε, κατόγουν ε, βάσει το, του είδους των ιδίων πόρων, ε, το, βάσει της αρχής της μεταφοράς κονδυλίων ανάμεσα στα διάφορα ταμεία και σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται προ το παρόν οι ανησυχίε του Κοινοβουλίου και πιο συγκεκριμένα τη Επιτροπή των Μεταφορών. Πάντω, η έκθεση του Μαριάν νομίζω ανταποκρίνεται στι πραγματικέ μα ανάγκε και σίγουρα θα τύχει ε, υποστήριξη από όλου. Ευχαριστούμε, Μάριαν Κιλίν. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρινέσκου. Είναι εξαιρετικό το έγγραφο εργασία που υπέβαλε. Οι σκιώδεις εισηγητές ήταν σχετικά ομόθυμοι ως προς το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης. Δέκα δίσε χρησιμοποιούμε κάθε στιγμή ε, για την υποστήριξη των δικτών ε, καυσίμων. Ε, με τέτοια ποσά θα πρέπει να συνειδητοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι χρειαζόμαστε τα κονδύλια μας για να χρηματοδοτήσουμε και την βιώσιμη ανάπτυξη. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τα περιβαλλοντικά έργα θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλητα και η χρηματοδότηση θα πρέπει να αποσκοπεί στην μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και ε, άλλες ε, δυσμενείς επιπτώσεις ε, για το περιβάλλον. Επίσης είναι σημαντικό η στόχη μας για τη χρηματοδότηση να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις όλων των εμπλεκομένων φορέων. Δυστυχώ ε, δεν έχει επικρατήσει διαφάνεια ω προς ε, τα αιτήματα του τομέα των μεταφορών για τη χρηματοδότηση, να θυμηθούμε, παραδείγματο χάρη, πώς ε, έχουν διοχετευτεί τα κονδύλια σε λιμένες όπου δεν βγαίνουν τα πλοία ή σε αερολιμένες όπου δεν προσγειώνονται αεροπλάνα. Θα πρέπει να τονίσω επίσης πως εχουν διοικητευτεί τα κονδυλια σε λιμενες οπου δεν βγαινουν τα πλοια η σε αερολιμενες οπου δεν προσγειωνονται αεροπλανα θα πρεπει να τονισω επισης πως χρειάζεται άμεση αντίδραση από πλευράς μας για να προστατεύσουμε τον τομέα των μεταφορών και να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας γύρω από την υποδομή, διότι οι υποδομές που διαθέτουμε δεν επαρκούν. Δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε σε υδροδρομικά δίκτυα, από μόνο του δεν εξυπηρετούν τι ανάγκε μα. Θα χρειαστούμε μια αποτελεσματικότερη χρήση του δυναμικού που υπάρχει και να το συνδυάσουμε με αναδιαμόρφωση του συστήματο μεταφορών. Μόνο έτσι θα έχουμε σοβαρέ πιθανότητε να στοχεύσουμε τα προϊόντα και τι υπηρεσίε που βασίζονται στην αποτελεσματική χρήση των ε, οχημάτων και των υποδομών. Πρόκειται για μια μεγάλη αλλαγή και θα ήθελα να ε, ζητήσω την υποστήριξη για την τροπολογία 62. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Καρή Μαντέλη, παρακαλώ. Πρόεδρε. κυρία Ντελή, ευχαριστώ. Από την ομάδα των οικολόγων έχουμε υποβάλει διάφορες τροπολογίες ε, και μα ικανοποιεί το γεγονό ότι ενσωματώθηκαν κάποιε από αυτέ. Ε, η τροπολογία μα επί του μακροπεριφερειακού ε, συντονισμού για τα διασυνοριακά επίσης μας βρίσκει ικανοποιημένο, αλλά υπάρχουν δύο σημεία που θα θέλαμε να σχολιάσουμε. Καταρχάς, κάτι αρκετά σοβαρό. Είναι η απουσία οποιασδήποτε εκτίμησης της COP21. Εδώ είμαστε σε ένα πλαίσιο αναθεώρηση του πολιετού δημοσιονομικού, από την άλλη όχι τόσο κλασικό, γιατί βεβαίω ε, ο πραγματικός σεισμός ο πολιτικός ήταν η Συμφωνία του Παρισίου. Πέρα από την ε, Κομισιόν Γιουνκέρ που τον υποστήριξε Άρα υπάρχει ένα στοιχείο που λείπει και που η Επιτροπή μας θα πρέπει να το έχει υπόψη της κάθε φορά που εξετάζει μία έκθεση δημοσιονομική ή έκθεση 2007-20 που θα είναι απόρρια των συμφωνιών του Παρισιού. Και επομένως τα κράτη-μέλη θα κληθούν να την εφαρμόσουν τη συμφωνία αυτή. Και θα θέλαμε σε αυτήν την έκθεση δημοσιονομική να το βλέπουμε αυτό. Για να βλέπουμε και την ε, συμμόρφωση προς την COP21, προς τη μείωση των εκπομπών. Και αυτή είναι ακριβώς η έννοια της τοπολογίας 4 που υποβάλαμε. Και ελπίζουμε ότι θα εγκριθεί. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Τα μεγάλης κλίμακος έργα Ο εισηγητής απέρριψε την τροπολογία μας. Δεν πάβουν οι διαμαρτυρίες, ειδικά σε ένα πλαίσιο CF, σχετικά με την απουσία τέτοιου είδους έργων. Δεν κατανοώ γιατί όταν μιλούμε για μεγάλα έργα έχουμε ένα οντολογικό θα έλεγα πρόβλημα διότι έχουμε ε, καταναλωτές χώρου οικονομικών υπηρεσιών πόρων και εστιαζόμαστε τελικά σε έργα μικρότερης κλίμακας που έχουν όμως πολύ μεγαλύτερη αξία για την βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη. Πρέπει να εξασφαλίσουμε εδώ δηλαδή ότι έχουμε λάβει, ότι μάλλον διαβιβάζουμε το σωστό μήνυμα προς την Κομισιόν σχετικά με τη βελτίωση των υφισταμένων υποδομών. Το δεύτερο θέμα είναι το θέμα της διαφάνειας. Είναι απαράδεκτο και δεν είναι και επικοδομητικό να μην έχουμε διαφάνεια σε ένα έργο της γραμμής του Τωρίνου όπως είναι αυτή, δηλαδή αυτό το έργο, γιατί πρέπει να το πούμε, δεν έχουμε τους πόρους. Αυτή η, κλίση, η έκκληση για διαφάνεια είναι κάτι που το συμμερίστηκαν όλες οι πολιτικές ομάδες. Κατά τα λοιπά, δεν μπορώ παρά να χαιρετήσω την εξαιρετική δουλειά του κυρίου Μαρινέσκου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Γεώργη Πυρίνσκη ο επόμενος, παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη βέβαια για το ότι δεν ήμουν προηγούμενα έγκαιρα παρόν στην έναρξη της συνεδρίασης. Θα ήθελα, ωστόσο, να προσθέσω τη φωνή μου, εκφράζοντας και εγώ την εκτίμησή μου για το έργο που επιτελέστηκε από τον κύριο Μαρινέσκου. Και όσον αφορά τις αρχικές του προτάσεις, που αποδείχθηκαν ότι θεμελιώνονται με πολύ καλό τρόπο, σε πολύ καλή βάση, θεσπίζοντας τις κυριότερες προτεραιότητες στις οποίες θα πρέπει να εστιαστεί και να δώσει συνέχεια στο μέλλον η κοινοβουλευτική μας επιτροπή σε σχέση με την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου και αυτό καταδεικνύεται και στους συμβιβασμούς που επετέφθησαν. 11 ή 12 συμβιβασμοί που υποστηρίζονται από ένα μεγάλο εύρος, ένα μεγάλο φάσμα πολιτικών κοινοβουλευτικών ομάδων. Και είναι σημαντικό να το πούμε ότι αυτές οι συμβαστικές προτάσεις περαιτέρω αναπτύσσουν τις αρχικές θέσεις που είχαν εκτεθεί, είχαν προταθεί. Δύο-τρία θέματα θέλω να τονίσω. Ένα, το οποίο αναφέρει ο κύριος Μαρινέσκου, πιστεύω στην αρχή της ε, παρουσίασης το, το έθεσε, ότι είναι σημαντικό όχι μόνο να επιχειρηματολογήσουμε ότι χρειαζόμαστε πρόσθετα κονδύλια, και για την ε, επαναχρησιμοποίηση ε, και για την, ε, τα σχέδια τα ευρωπαϊκά τα οποία πρέπει να χρηματοδοτηθούν αλλά επιπλέον και για την υλοποίηση, εφαρμογή του προϋπολογισμού και το συντονισμό μεταξύ των διαφορετικών προτεραιοτήτων πολιτικής. Να τονίσουμε τις στρατηγικές μας για τις περιφέρειες που πρέπει να τονιστούν και πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, διότι αυτό πιστεύω πάλι ότι στοχεύει στην ίδια κατεύθυνση όπως και κάποιοι από τους συμβιβασμούς, δηλαδή να τονίσουμε τη σπουδαιότητα της συνοχής για την οποία συνοχή και οι μεταφορές και ο τουρισμός διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Κάτι που βρίσκεται στον πυρήνα, στην καρδιά της πρόκλησης των προκλήσεων που αντιμετωπίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα και τα οποία όλα αυτά σχετίζονται ιδιαίτερα με την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αυτών σχεδίων. Δεν θέλω να αναλώσω περισσότερο από το χρόνο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Έχουμε ισχυρή τοποθέτηση και θέση και πρέπει να ενωθούμε ώστε να την υπερασπιστούμε σε σχέση με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για την Επιτροπή τώρα παρακαλώ, ο κύριος Στεφανουάκη θα λάβει τον λόγο. Thank Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Για, αυτή, για αυτές τις τροπολογίες και τη συζήτηση θα ήθελα να περιοριστώ όμως στη διευκρίνηση κάποιων που σχετίζονται με την νομική πτυχή του ΣΕΦ. Προτείνεται εδώ ενθαρρύνεται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, κάνει, να αναλάβει κάποια δράση σε σχέση με το κονδύλιο της συνοχής του ΣΕΦ. Τι σημαίνει αυτό μετά τη 31η Δεκεμβρίου του 2016. Οποιαδήποτε κονδύλια δεν έχουν χρησιμοποιηθεί θα διέπονται από τον κανονισμό αυτό και θα χρησιμοποιούνται χωρίς να γίνονται σεβαστές οι, τα, οι εθνικές προσθέσεις, τα εθνικά κονδύλια που είχε προαποφασίσει για τα έτη 2014, 2015 και 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε εκτός και αν η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση και επιτρέψουμε στη διαδικασία συναπόφασης για την τροποποίηση αυτών των διατάξεων. Αλλιώς δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκταμιεύσει αυτά τα κονδύλια εκτός των κρατών μελών. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν αυτό, διότι ε, προορίζονται αυτά τα κονδύλια για τα κράτη συνοχής. Πρώτον και δεύτερον, δεν θα είναι δυνατόν ή ούτε να παρατείνουμε αυτή την περίοδο εθνικών κονδυλίων πέραν από την περίοδο που αναφέρεται στον ίδιο τον κανονισμό, ούτε και γίνεται να επαναειραρχήσουμε με συγκεκριμένο τρόπο τις προτεραιότητε, αποκλίνοντα έτσι από τι διατάξει του κανονισμού για το ΣΕΦΕ, διότι για την υποστήριξη μέσω επιδοτήσεων και κυρίω για το κονδύλι συνοχή, έχουν ήδη ιεραρχηθεί οι προτεραιότητε. Αυτά τα δύο ήθελα να τα διευκρινίσω, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα μπορέσει να δώσει αλλιώ συνέχεια στα αιτήματά σα. Και κάτι άλλο που νομίζω έχει μια βαρύτητα σε σχέση με τον αριθμό τροπολογιών που αναφέρονται σε αυτό είναι το θέμα τη συνολική διαχείριση των ε, επιλέξιπων προγραμμάτων ε, στην πρώτη και δεύτερη υποβολή ε, προτάσεων πρόταση υποβολή προσφορών. Και στα πλαίσια του, ε, της δεύτερης πρότασης ε, υποβολής έχουμε το use it or lose it. Είναι αυτή η αρχή του χρησιμοποιήστε τα κονδύλια ή χάστε τα. Δηλαδή ε, έχουμε την επιλογή των ε, προγραμμάτων και στη συνέχεια περιμένουμε την εφαρμογή. Όταν όμως καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι είναι πολύ σημαντική η καθυστέρηση ή κα, καταργούνται τα προγράμματα ή ακυρώνονται, η καταργουνται τα προγραμματα πρακτική είναι να περιορίσουμε τη χρηματοδότηση για αυτό το πρόγραμμα ή να την ακυρώσουμε ως δί να επαναδιοχετεύσουμε τα εξοικονομηθέντα κονδύλια ε, στο Ταμείο για να χρηματοδοτηθούν περαιτέρω δράσεις. Η Επίτροπος ε, Μπούλτς ε, φυσικά θα σας εξηγήσει ποιο είναι το όραμά για τους μελλοντικούς διαγωνισμούς που θα γίνουν. Σε αυτό το πλαίσιο όμως υπάρχει μια σημαντική ευελιξία έμφυτη μέσα στο σύστημα ούτως ώστε ε, τα διαθέσιμα κονδύλια ε, στα πλαίσια του ΣΕΦ να χρησιμοποιηθούν γιατί ήδη ε, έχουν διοχετευτεί, θα διοχετευτούν σε συγκεκριμένα διαρθρωτικά προγράμματα και έχουμε αυτή την ευελιξία λοιπόν ή χρησιμοποιούνται τα κονδύλια από ένα πρόγραμμα ή τα χάνουν οι δικαιού και χρησιμοποιούνται για άλλα πρόγραμματα. Ευχαριστούμε και πάλι ο εισηγητής τώρα ο Μαριάν Μαρινέσκου. President. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και πάλι τους συναδέλφους για τα καλά τους λόγια και την ε, στήριξη. Αναφερόμασταν σε μια τροπολογία σε ένα συγκεκριμένο έργο, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και ζητώ συγγνώμη. Η αναθεώρηση ζητείται από το ίδιο το MFF. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη μνήμα στην COP21 η αναφορά στα πορίσματα της σημαντικής αυτής συνάντησης υπάρχει. Για τα σχόλια της Κομισιόν φυσικά και δεν μπορεί να κάνει η Κομισιόν κάτι που δεν προβλέπει διάταξη του κανονισμού έχουμε ζητήσει τροποποιήσεις και θα δούμε κατά πόσο η μεταρρύθμιση θα πηγαίνει και στους βασικούς κανονισμούς. Εμείς είχαμε ζητήσει περισσότερους πόρους, είχαμε ζητήσει προέκταση της προθεσμίας για τους, τα κονδύλια συνοχής και είχαμε ζητήσει να χρησιμοποιούνται τα κονδύλια αυτά για συνοριακά έργα που συμπεριλαμβάνονται ήδη στο παράρτημα του ΣΥΕΦ. Είναι επομένω ε, σαφέ ότι είναι συγκεκριμένο αυτό στο οποίο αναφερόμαστε εδώ. Σα σας ευχαριστούμε. Το πρώτο σημείο λοιπόν ολοκληρώθηκε. Θα ψηφιστεί αύριο το απόγευμα κατ' εξαίρεση. Τις έχουμε τρίτη πρωί τις ψηφοφορίες. Αύριο το απόγευμα κατ' εξαίρεση θα ψηφίσουμε για αυτή την έκθεση κατ' εξαίρεση. Και μια και δεν μπορεί να προσέλθει νωρίτερα η Επίτροπος για το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, θα διακόψω τη συνεδρίασή μας. Και στις 4 θα συνεχίσουμε, εντάξει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μετά από αυτό το σύντομο διάλειμμα μπορούμε να συνεχίσουμε με τη συνεδρίασή μας. Ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο Βιολέτα Μπούλτς για το πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπο, Επιτροπής όσον αφορά το εφσι για τα προγράμματα και σχέδια μεταφορών. Σας καλοχαιρετίζουμε, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Η σημερινή ανταλλαγή απόψεων διεξάγεται μέσα στο διαθρωμένο διάλογο και εξυπηρετεί το στόχο να εξετάσουμε την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2016 και την προπαρασκευή για το πρόγραμμα εργασίας για το έτος 2017, λαμβάνοντας υπόψη πάντα φυσικά τις αποφάσεις ε, που ελήφθησαν πέρυσι και σε σχέση με το ΕΦΣΙ και ΣΕΦ και την υποστήριξη σε σχέση με τα κονδύλια. Κυρία Βιολέτα Μπούλτς, έχετε τον λόγο. Παρακαλώ. Thank you very much. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχαήλ. Αγαπητοί συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου προσφέρετε να μιλήσω για αυτό το σημαντικό πραγματικά εγχείρημα, το σημαντικό θέμα, ιδιαίτερα για τις επόμενες εβδομάδες. Ε, βρίσκομαι εδώ όπως ο Μιχαήλ προανέφερε ώστε να σας προσφωνήσω και να σας μιλήσω για τους μηχανισμούς διασύνδεσης ε, της Ευρώπης, το πρόγραμμα επενδύσεων του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Juncker, ιδιαίτερα για τους άξονες και πυλώνες για το ΕΦΣΥ, και για να σας ενημερώσω για τον ορίζοντα 2020 όσον αφορά τον τομέα των μεταφορών. Ωραία λοιπόν. Πρώτα απ' όλα να θέσουμε το πλαίσιο για τη συζήτηση όσον αφορά τις επενδύσεις αυτές και τους μηχανισμούς, επενδυτικούς μηχανισμούς. Να βεβαιωθούμε ότι γίνεται κατανοητό το όραμα μας και υπάρχει απόλυτη σαφήνεια για το, την επικέντρωσή μας, τον εστιασμό μας εστιαζόμαστε στην εσωτερική αγορά κυρίως, όπου θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, την άρση των προσκομμάτων και εμποδίων όσον αφορά την, ε, τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών που πρέπει να λειτουργεί καλά και συνολικά επικεντρωνόμαστε στην διασυνδεσιμότητα και την διευκόλυνση ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια και έχει έναν κυριότερο στόχο που έχει θέσει στις προτεραιότητές της ως στόχους, ε, την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος. Φυσικά αυτά μπορούν να επιτευχθούν ε, μέσω απόλυτης αφήνειας της ψηφιοποίησης ε, του συντονισμού με στοχοθετημένες λύσεις, ε, παγκοσμιοποιημένες ε, στοχεύσεις και υποστήριξη όσον αφορά την καινοτομία και τις επενδύσεις. Είναι σαφέστατο λοιπόν οτιδήποτε πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να διαρωτόμαστε επικεντρωνόμαστε σε αυτές τις κύριες προτεραιότητες και στρατηγικές που θέλουμε να υλοποιήσουμε ή όχι. Φυσικά θα επικεντρωθούμε στις επενδύσεις σήμερα σαν έναν από τους μηχανισμούς που θα προωθήσουν αυτό, αυτά τα σχέδια. Είναι βέβαιο ότι τους επόμενους μήνες θα συζητήσουμε και άλλα θέματα, την ψηφιοποίηση για παράδειγμα και ούτω καθεξής. Επενδύσεις. Γιατί να υπάρξουν επενδύσεις. Για να μπορέσει η Ευρώπη να ανταποκριθεί σε αυτές τις προτεραιότητες πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις. Αν δεν υπάρξουν επενδύσεις δεν θα υπάρξει ανάπτυξη. Αν δεν υπάρξει ανάπτυξη δεν θα μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο. Λοιπόν, να υπάρχει διασύνδεση αραγής και συνεχής να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των καταναλωτών, των πολιτών καταναλωτών αφενός και επιχειρηματιών και επιχειρήσεων, ώστε η Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική και να είναι αποτελεσματική. Ένα από τα κυριότερα θέματα λοιπόν είναι να μπορέσουμε στην παγκοσμιοποίηση να διασφαλίσουμε να είμαστε εμείς να έχουμε ρόλο προπομπού, πρωτοπόρου σε όλα αυτά. Για να μπορέσουμε να τα πετύχουμε αυτά <clears throat> είναι δύο στοιχεία απόλυτα απαραίτητα έρευνα και καινοτομία αφενός που έτσι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέα μέσα, νέα εργαλεία τεχνολογικά όσον αφορά την τεχνολογία αλλά και την κοινωνία, κοινωνικά, κοινωνικές ανάγκες. Εδώ θέλω να τονίσω την ανάγκη του αναδυόμενου προτύπου των στήτ ε, ε, δημοσίων ε, και ιδιωτικών συνεργασιών και σε αυτό θα στραφούμε και όσον αφορά την επόμενη παρέμβαση. Να δούμε τι έχει γίνει μέχρι σήμερα για την βελτίωση των επενδύσεων στις μεταφορές. Ποιοι μηχανισμοί υπάρχουν ώστε να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί σε επενδύσεις. Θα επικεντρωθώ λοιπόν σε τρία. ΣΕΦ, είναι ο πυρήνας ε, των μηχανισμών, διαθροτικά ταμεία, εδώ επικεντρωνόμαστε κυρίως στην περιφερειακή ανάπτυξη και το ΕΦΣΥ το έτσι ε, και που πραγματικά υπόσχεται πάρα πολλά και είναι ένας μηχανισμός που μπορεί να δώσει όχι μόνο προσδοκίες αλλά να υπάρξουν και αποτελέσματα για πρόσθετη χρηματοδότηση. Για τον τομέα των ε, μεταφορών και των υποδομών και τις επενδύσεις άμεσα, τα κράτη-μέλη με τους ε, επιμέρους μηχανισμούς ε, που προβλέπονται και τα άλλα θεσμικά όργανα με τους μηχανισμούς τους πολλά έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Όμως θα ήθελα να επικεντρωθούμε σε αυτά που έχει άμεση επιρροή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που σε αυτά επικεντρωνόμαστε κυριότερα στις δραστηριότητες μας. Ας αρχίσουμε πρώτα με το ΣΕΦ. Έχουμε λοιπόν εδώ την ανάγκη του να υπάρξει η ενδυνάμωση της ραχοκοκαλιάς της οικονομίας μας. Θα συνεχίσουμε με τις προσπάθειές μας για να μπορέσουμε μέχρι το 2030 να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο για τους διαδρόμους. 700 δις περίπου ευρώ επενδύσεων έχουν ταυτοποιηθεί και εντοπιστεί. Οι ανάγκες για πάνω από 700 δις ευρώ είναι τεράστιο ποσό αυτό και επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι έχουμε σε αυτή την εντολή τον μεγαλύτερο οποτεδήποτε προϋπολογισμό για τις μεταφορές. Αν δούμε αυτό τον όγκο, υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ αυτών που είναι διαθέσιμα τα, ως κονδύλια και αυτών που πρέπει να διασφαλιστούν επιπλέον. Πρέπει να γίνει αυτό, να διασφαλιστούν. Αλλά να δούμε τι κατάφερε το ΣΕΦ μέχρι σήμερα. Πρώτα, με έναν προϋπολογισμό 12,77 δις ευρώ από το 2014 και μέχρι το 2015 δόθηκαν σε 263 προγράμματα κονδύλια του ΣΕΦ και είχαμε 28,83 δις, δισεκατομμύρια επενδύσεων. Αυτά με την πρώτη αυτή, με την πρώτη προσπάθεια, τον πρώτο γύρο. Ταυτόχρονα είχαμε και τριπλάσιο όγκο που μπόρεσε να δημιουργηθεί. Υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες εδώ. Πολλά προγράμματα και σχέδια που πρέπει να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν πρέπει να διασφαλίσουν τα κονδύλια αυτά. Υπό την σημερινή λοιπόν πραγματικότητα 427 έργα έχουν υποβληθεί <clears throat> με τον συνολικό όγκο που συνεπάγονται, δηλαδή διπλάσιο όγκο από εκείνον που είχε προβλεφθεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι και σε αυτό το πεδίο έχουμε και την δυνατότητα της ψηφιοποίησης και των ευφυών ε, λύσεων. Στον τρίτο γύρο που μέχρι τα τέλη του 2016 θα πρέπει να ολοκληρωθεί και μέχρι το 2018 θα έχουμε τις ε, υπόλοιπες δράσεις για όσα συνέβησαν μέχρι σήμερα από πλευρά ΣΕΦΑ βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντικά. Ο δεύτερος μηχανισμός που θέλω να εποπτεύσουμε τάχει είναι ο ορίζοντας 2020. Η επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Το 2014 είχαμε 517 ε, εκατομμύρια ευρώ τήθηκαν στη συνέχεια επιπλέον 219 ε, εκατομμύρια ευρώ. Για το 2016 επιπρόσθετα 434 εκατομμύρια ευρώ θα είναι αναγκαία να διατεθούν για την ε, χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη γεφυροποίηση του χάσματος μεταξύ της ε, έρευνας και των δυνατοτήτων απασχόλησης καινούριο το 2016-2017 θα είναι κέντρο βάρους ε, ο αυτοματισμός. 3,5 εκατομμύρια ευρώ για την ε, αναπτύξη των καθαρών κινητήρων. Επίσης ε, αποκοινούμε τα κοινά εγχειρήματα για τις μεταφορές και την δυνατότητα να καλυφθούν άλλα χαρτοφυλάκια όσον αφορά το, την χρήση του υδρογόνου συνολικά 2,7 δις θα είναι ο προϋπολογισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το πρόγραμμα. 3 δις τουλάχιστον ευρώ στις περαιτέρω συνεισφορές και παρεμβάσεις από τις βιομηχανίες θα πρέπει να διασφαλιστούν ώστε να είμαστε καθαροί και αποτελεσματικοί όσον αφορά τις, ε, τους πόρους μας, ε, τις υποδομές, ε, τις υπηρεσίες και ταυτόχρονα να βελτιωθεί η κινητικότητα και να βελτιωθούν και οι μεταφορές στα αστικά κέντρα, στις αστικές περιοχές. Με πολύ στοχοθετημένο και αποτελεσματικό τρόπο λοιπόν ενεργούμε. Περνάμε στο επόμενο πρόγραμμα τώρα για την Ευρώπη από πλευράς ΕΦΣΗ Όπως γνωρίζετε <clears throat> έχουμε τρεις κύριους πυλώνες που υποστηρίζουν αυτό το πρόγραμμα. Ένας πυλώνας ε, αφορά το, τις επενδύσεις που θα είναι πιο προβλέψιμες και συνδέονται με τα ε, ρυθμιστικά πλαίσια τα οποία είναι αναγκαία ώστε από πλευράς κρατών μελών να είναι διαφανή αυτά τα πλαίσια και να είναι προβλέψιμες οι εξελίξεις όσον αφορά τους επενδυτές. Να υπάρχει μια σταθερότητα ακόμα και αν υπάρχει αλλαγή κυβερνήσεως σε κάποια χώρα να είναι όλα προβλέψιμα και σε ένα σταθερότερο πλαίσιο. Δεύτερος πυλώνας είναι ένας πολύ σημαντικός στην τεχνική υποστήριξη πυλώνας. Στις προηγούμενες προσπάθειές μας αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει απουσία τεχνικής υποστήριξης για τέτοιου είδους δράσεις. Γι' αυτό λοιπόν αυτός ο δεύτερος πυλώνας ε, εστιάζεται ισχυρότερα, εντονότερα στην τεχνική υποστήριξη και την συμβουλευτική δράση για την ε, αρρωγή των ε, επενδυτών όσον αφορά τα εγχειρήματα αυτά. Οι μεταφορές είναι ο δεύτερος πιο δημοφιλής τομέας για την υποβολή τέτοιων προτάσεων μέσα σε, από αυτό το κέντρο. Μέσα στο κέντρο, από το κέντρο αυτό θα θέλαμε να είμαστε πιο ενεργοί στην προσέγγισή μας. Το hub αυτό θα υποστηρίζει τις εξελίξεις ώστε να υπάρχει η ενδυνάμωση δυνατοτήτων από πλευράς των κρατών μελών και επιχειρηματιών οι ε, μεταφορές που χρησιμοποιούν αυτά τα κονδύλια εντονών ανώτερα και προγράμματα και ε, δράσεις που πρέπει να προετοιμαστούν για τις ε, ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν διαφορετική κλίμακα και διαφορετική ένταση. Αυτό είναι ο κομβικός τομέας στον οποίο πρέπει να, πρέπει να μπορέσουμε να συντονιστούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει η υλοποίηση όλων αυτών να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Στοχοθετημένη τέτοια προσέγγιση θα είναι απόλυτα αναγκαία στο μέλλον. Επιπρόσθετα είναι κέρια σημασία ε, το ΕΦΣΙ να είναι αποτελεσματικό σε όλα τα κράτη-μέλη. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το ΕΦΣΙ θα μπορέσει να καλύψει τις, ε, τα χάσματα και τι διαφορές μεταξύ Ανατολής και δύση. Αυτά τα πρώτα αποτελέσματα σε αυτή την πρώτη φάση δεν στοχεύουν προς αυτή την κατεύθυνση της γεφυροποίησης δηλαδή και της κάλυψης των διαφορών. Από όλα τα προγράμματα που βρίσκονται υπό εξέλιξη, μόνο ένα είναι ε, αυτό το οποίο αφορά την συνοχή και αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις διαφορές γιατί διαφορετικά θα υπάρξει ένα μεγάλο χάσμα στην ανάπτυξη μεταξύ της Δύσης, των χωρών της Δύσης και της Ανατολής. Και γι' αυτό στην ε, ε, Υπουργική Συνάντηση και με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων 22 Απριλίου στην Λιουμπλιάνα όπου ήταν παρόντες ε, και παρούσες αντιπροσωπείες και αντιπρόσωποι για να ε, συνειδητοποιήσουμε το τι μπορεί να χαθεί αν δεν εμπλακούμε στην χρήση των νέων μηχανισμών και συντονιστικών μέσων, αλλά ταυτόχρονα αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει έλλειψη γνώσης, τεχνογνωσίας, πραγματογνωμοσύνης, ιδιαίτερα στον τομέα των ε, ε, οικονομικών και των ε, τεχνικών οικονομικών των ρυθμίσεων. Τώρα, περνώ στο εύση και την διευκόλυνση ρευστότητας και κονδυλίων στην αγορά και για πιο στοχευμένη χρήση των κονδυλίων. Είναι ισχυρή η συνιστόσα του ΕΦΣΥ, 12,8 δις ε, ευρώ για τα προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν <clears throat> και ένα όγκο συνολικό 100 δις ευρώ. Από το Διευθυντικό ε, Συμβούλιο έχουν εγκριθεί τέτοια προγράμματα και ευελπιστώ ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να τα εγκρίνουμε όλα παραδείγματα. Πλατφόρμα για την ε, ε, επιτάχυνση επενδύσεων όσον αφορά τις ε, λιμενικές υπηρεσίες και τους λιμένες στην Ισπανία, προγράμματα υποδομών στην Ιταλία και την διάθεση όλων αυτών των δυνατοτήτων τεχνογνωσίας. Αυτά τα έργα μεταφορών έχουν το δυναμικό να δημιουργήσουν περίπου 60.000 θέσεις απασχόλησης τα επόμενα έτη είναι κατεκτήμηση είναι αυτό και είναι προσωρινής απασχόλησης εργασίες, ε, έργα και θα πρέπει να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε σε πιο μακροχρόνιο πλαίσιο, με ένα πιο μακροχρόνιο ορίζοντα, ώστε να μπορέσουν τα δισεκατομμύρια αυτά επενδύσεων να μπορέσουν ταχύτατα να διατεθούν επιτρέποντας ε, την εκτίμηση ότι περίπου πάνω από 500.000 θέσεις απασχόλησης θα μπορέσουν ε, να διατηρηθούν στο εγγύς μέλλον. Το δυναμικό είναι ισχυρό Πολύ ισχυρό λοιπόν και παράλληλα θα πρέπει ε, να δούμε τον συνολικό όγκο για το 2015 που ήταν 12,5 ε, δις. Ε, ε, είχαμε πρόσφατα την ανακοίνωση από πλευράς των ηθινόντων ότι θα διατεθούν επιπρόσθετα 4,5 δις ευρώ με το νέο τερματικό σταθμό 3 του αεροδρομίου της Φραγκφούρτης νέα τρένα όσο όσον αφορά το ε, δίκτυο του ε, Λίβερπουλ. Δεν θα πρέπει όμως να πούμε ότι μας ικανοποιούν όλα αυτά και εφησυχάζουμε Δεν μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώθηκε το έργο μας και έτσι μπορούμε να εφησυχάσουμε πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα μιας ε, ενδυνάμωσης που θα δώσει την δυνατότητα να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης δίνοντας τη δυνατότητα στους πλειοκτήτες να χρησιμοποιούν ε, πιο καθαρούς ε, κινητήρες στα πλοία τους ώστε να επιβαρύνεται λιγότερο το περιβάλλον από εκπομπές ρήπων. Επίσης όσον αφορά τους σιδηροδρόμους ε, και τις αερομεταφορές επενδύσεις σε πλατφόρμες ώστε να μπορέσουν σε μικρότερες πλατφόρμες να διασφαλιστούν οι επενδύσεις με καθαρά οχήματα. Προωθούμε μια καλή αποτελεσματική λύση για πολυεθνικά προγράμματα. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα εκπονηθεί ένα μέσο, ένα εργαλείο από πλευράς μας για ένα πρόγραμμα επενδύσεων που μπορεί να δώσει την δυνατότητα να μπορούν παραγγελίες από οπουδήποτε στην Ευρώπη για ηλεκτρικά λεωφορεία για παράδειγμα να μπορέσουν να λειτουργήσουν, να μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις από κράτη ε, και να μπορούν από τους παρόχους ε, ή τους, ε, τις διάφορες βιομηχανίες να διατίθενται αυτά τα αναγκαία οχήματα ή μέσα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δυναμικό για το, για το μέλλον. Όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτά τα σχέδια επενδύσεων θα πρέπει να ενδιαφέρονται άμεσα στην καινοτομία και μέχρι σήμερα έχουμε καλή, ας το πω έτσι, ανταπόκριση από τους ενδιαφερόμενους. Πρέπει να πω ότι έχουμε σημειώσει πρόοδο σε σχέση με πέρσι, αλλά έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε και ε, είχαμε ε, ε, ενεργό υποστήριξη σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε να είναι στοχευμένη η υποστήριξη που προσφέρουμε σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους με ομοιόμορφο τρόπο σε, στα 28 κράτη-μέλη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας παρακαλώ να το περάσετε και εσείς στις εκλογικές σας περιφέρειες αυτό το μήνυμα. Μιλήστε στις χώρες σας, στους πολίτε. Ε, για να συμμετάσχει σε αυτή την εκστρατεία ευαισθητοποίησης για να υπάρξει καλύτερη κατανόηση των νέων ε, ε, χρηματοπιστωτικών εργαλείων, διότι για να έχουμε μεγάλη, μεγαλύτερη πρόοδο θα χρειαστούμε αυτό το περίφημο το blending, δηλαδή ε, συνδυασμό επιδοτήσεων και δανείων. και θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τις ικανότητες μας χρήση αυτών των μηχανισμών. Τι έπεται πρώτον το επενδυτικό πρόγραμμα για την Ευρώπη, για το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα στον τομέα των μεταφορών. Και ζητώ την υποστήριξή σα, τη χρειάζομαι, αλλά υπάρχει ένα πελώριο ανεκμετάλλευτο δυναμικό. Είμαι αισιοδόξη, όμω θα πρέπει και εμεί να κάνουμε το κομμάτι που μα αναλογεί. Για να τα καταφέρουμε, πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε ένα στρατηγικό πρόγραμμα, ώστε να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη και τους προμότερους των προγραμμάτων για τη μετάβαση από τις, ε, την προσέγγιση της ε, κρατικής χρηματοδότησης προς τη χρήση των νέων χρηματοπιστωτικών μηχανισμών. Εδώ σας μιλάω για νέα κουλτούρα, νέα προσέγγιση στον τομέα των μεταφορών και ξέρετε πως εσείς ξέρετε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να αλλάξουν οι συνήθειες, όμως κάποιος πρέπει να το κάνει. Γιατί όχι εμείς. Ναι. So, no matter what, uh, Όπως και να έχει, πέρα από τις επιδοτήσεις χρειαζόμαστε αυτό το blending, όπως λέγαμε, το συνδυασμό με τα δάνεια. Αυτό μας ε, ε, βοηθάει να αντιμετωπίσουμε το χρηματοδοτικό ε, κενό, ενώ λειτουργεί ως καταλήτης για τις επενδύσεις το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Θα ήθελα λοιπόν να ακολουθήσουμε μια πρακτική προσέγγιση. Αυτή η διαδικασία blending επιδοτήσεων και δανείων χρησιμοποιήθηκε στο Δουβλίνο, στο Καλέ, στα βασικά λιμάνια δηλαδή και στο ΣΕΦ, ε, στο Μηχανισμό Συνδέοντα στην Ευρώπη και θα χρησιμοποιηθεί για τα προγράμματα έτσι στην Σλοβακία όπω σα έλεγα προηγουμένω και γενικότερα στο πλαίσιο του ΣΕΦ, ε, του Συνδέοντα στην Ευρώπη ε, γιατί τώρα γίνεται και αξιολόγηση και σίγουρα θα βρεθούν νέα ενδιαφέροντα προγράμματα που θα είναι κατάλληλα για τη διαδικασία blending, όχι μόνο για επιδοτήσεις δηλαδή. Λοιπόν, για τις επιδοτήσεις ΣΕΦ νομίζω ότι έχουμε πολύ ισχυρή επιχειρηματολογία, γιατί στο επόμενο πολιετές μετά την αναθεώρηση θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα κονδύλια που κατά προτεραιότητα χρησιμοποιηθούν για υποστηριχθεί αυτή η νέα διαδικασία blending. Εγώ θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια. Ό,τι περνάει από το χέρι μου θα το κάνω, όμως χρειάζομαι την βοήθειά σας. Ε, θα αγωνιστώ, θα πολεμήσω για τις μεταφορέ ε, διότι μπορεί πολλοί άλλοι να προσπαθήσουν να οικειοποιηθούν αυτά τα ελάχιστα επιπρόσθετα κονδύλια που θα καταστούν διαθέσιμα και είναι ξαναλέω ισχυρή επιχειρηματολογία μας. Και ξέρω ότι θα υπάρξει υποστήριξη, όμω και από πλευρά των πολιτικών χρειαζόμαστε υποστήριξη, αλλιώ δεν τα καταφέρουμε, αγαπητοί αξιότιμοι βουλευτέ. Ε, ε, ήρθε η στιγμή να δείξουμε ότι είμαστε σε θέση να προσφέρουμε πραγματική προστιθέμενη αξία, ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Από κοινού μπορούμε να σημειώσουμε ε, επιτυχία σε αυτόν τον νέο μα αγώνα. Θα ήθελα επίσης να σε επενθυμίσω και τις ημέρες TNT ε, στο Ρότερνταμ φέτος, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα δηλαδή. Είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της διάσκεψης για τους ε, επενδυτές ε, και για τους δικαιούχους. Θα κάνουμε speed dating ανάμεσα τους και θα σε συναντήσεις ανάμεσα στους επενδυτές και στους δικαιούχους που περιμένουν ναι, τις επενδύσεις, είναι έτοιμοι και επιλέξιμοι. Επίσης, επιπρόσθετο consulting, χρόνο δηλαδή που θα αφιερώσουμε στο consulting για τα προγράμματα που ακόμη δεν έχουν οριμάσει, όμως θα ήθελαν ε, να λάβουν κάποια πρώτα σχόλια. Αυτό θα γίνει με υποστήριξη από δικές μου υπηρεσίες ε, και Ε, με τους συντονιστές του διαδρόμου που θα είναι παρόντες επίσης ε, και τους ειδικού από την ε, ΕΤΕ. Ε, τρεις ποιοτικέ υπηρεσίες ε, που ε, ταυτόχρονα θα παραστούν στις ημέρες διευρωπαϊκών δικτύων τεντή, και έτσι θα έχουμε ολοκληρωμένη απόκριση όχι μόνο βάσει της παραδοσιακής προσέγγισης αλλά και από πλευράς επενδυτών και προμότερς των προγραμμάτων. Θα έχουμε τους δύο αντιπροέδρους, Κατάινεν και Σεύσοβιτς, θα έρθουν όπως και ο πρόεδρος της ΕΤΕ και ο αντιπρόεδρος και φυσικά όλοι εμείς. Οι θειασότες των μεταφορών. Ε, να είναι η αθρώη προσέλευση θα ήθελα να σας παρακαλέσω ούτω ώστε να σηματοδοτήσουμε αυτή τη νέα, το νέο σημαντικό στάδιο στην ε, εξέλιξη στον τομέα των μεταφορών. Ένα τελευταίο μήνυμα, κάτι άλλο που, πολύ σημαντικό που θα συμβεί στο Ρότερνταμ επίσης, ε, η δήλωση του Ρότερνταμ Ε, θα τονώσει τα βασικά δίκτυα μέχρι το 2030 για τα TNT και επίσης ε, καινοτόμα χρηματοδότηση για ε, την ΕΦΗ e και πράσινη υποδομή. Ελπίζω να προσέλκυσα και την προσοχή σας με, αυτά, με αυτή την παρουσίαση. Ελπίζω να σας δω στο Ρότερνταμ και κλείνοντας να επαναλάβω ότι πραγματικά βασίζομαι στην βοήθειά σας, στην ενεργού συμμετοχή σας. Ο, ο στόχος πραγματικά είναι να κατοχυρώσουμε τις βέλτιστες δυνατές ε, προϋποθέσεις ε, για να ε, φέρουμε την αλλαγή στον τομέα των μεταφορών. Σταματώ για να ακούσω τις ερωτήσεις, τα σχόλιά σας και φυσικά θα απαντήσω στη συνέχεια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Επίτροπε Βιολέτα Μπούλτς για όσα μας εκθέσατε. Περνάμε τώρα στη συζήτηση. Πρώτα ο κύριος Φαντέν παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ. Πέρυσι είχα πάει στις 10T ε, Days στη Ρίγα Και ελπίζω ότι η αντίστοιχη διοργάνωση στο Ρότερνταμ θα είναι εξίσου καλή. Γιατί αν είναι εξίσου καλή θα είναι τεράστια επιτυχία. Εγώ σε δύο ημέρες είχα συλλέξει πάρα πολλές πληροφορίες στη Ρίγα. Ελπίζω ότι θα έχουμε το ίδιο επίπεδο ενημέρωσης. Ένα άλλο σχόλιο όμως ήθελα να κάνω. Στην διάταξη αναφέρεται ότι σήμερα θα δούμε το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την εφαρμογή του για το 2016. Η Επίτροπος ανεφέρθηκε σε διάφορα μεγέθη για το CEF και το ΕΦΣΥ και οι συνάδελφοι, ιδιαίτερα ο κύριος Πίπα, θα επανέλθει στα μεγέθη αυτά αλλά ήθελα να ακούσω κάποια περισσότερα στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας της ε, Κομισιόν για το 2016. Όπως γνωρίζετε, το Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή προετοιμάζει τις παρατηρήσεις του σχετικά με το πρόγραμμα αυτό εργασίας το 2016 και θα ήθελα ιδιαίτερα να ακούσω κάποια πράγματα για το πακέτο των οδικών. Γιατί εκεί υπάρχει αρκετή ασάφεια θα έλεγα και δεν ξέρω αν θα μπορούσε η Επιτροπός ενδεχομένως να συντάξει ένα σύντομο έγγραφο για να μας εξηγεί το τι συνέβη. Γιατί αναφερθήκαμε στο πακέτο των οδικών αρχικά, μετά είχαμε σχόλια ότι προχωρούμε περισσότερο με την ε, διαδικασία της απαλλαγής από τον άνθρακα, αλλά όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και θα έχουν και σημαντικό αντίκτυπο κοινωνικό. Δεν ξέρω λοιπόν αν η Επιτρόπος Μπούλκ θα μπορούσε να μας πει κάποια περισσότερα πράγματα σχετικά με τις πολιτικές του 16 και τις προσδοκίες Κομισιόν για το 17. Γιατί υπάρχει σύγχυση και ασάφεια, επαναλαμβάνω. Και κυκλοφορούν, επιτρέψτε μου, και αρκετές ανοησίες. Άρα θα μπορούσε ίσως η Κομισιόν να μας πει περισσότερο για το παγιά των συνδεδρόμων, των οδικών, των αεροδρομικών, αλλά το συγκεκριμένο των οδικών δικτύων και η διασύνδεση του προγράμματος 16 με εκείνο 17 θα μπορούσε να είναι σίγουρα σαφέστερη. Αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Σέτσοκ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τα όσα μας εκθέσατε και την παρουσία σας. Παρουσίασή σας λέει κύριο Σέτουκ. Δύο-τρεις ερωτήσεις θα είχα που αφορούν τα ε, μελλοντικά τεκτενόμενα. Αναφερθήκατε στο 2030 που είναι έτος αναφοράς και έτος στο οποίο στοχεύουμε και θυμάμαι όταν ήμουν εισηγητή την τελευταία φορά από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια αναθεώρηση των δικτύων μεταφορών για το 2021-2022 είχε αναφερθεί. Διατηρείται αυτό, βρισκόμαστε εδώ σε σχέση με το σχεδιασμό κοντά στο σχεδιασμό και για τις ε, προσφορές ε, και για ε, ε, ε, τον επιμερισμό των έργων ήταν μία από τις προτεραιότητες της, του μηχανισμού σύνδεσης της Ευρώπης και των κατευθυντήριων γραμμών ότι θέλαμε διασυνοριακά τέτοια προγράμματα να προωθηθούν και αυτό είναι εκείνο το οποίο ας το πω έτσι κάπως με θλίβει το ότι τα κεντροανατολικά ευρωπαϊκά κράτη από πλευρά ζήτησης ε, δεν ήταν ιδιαίτερα ε, ενδυναμωμένα και αυτό ακριβώς το επιχείρημα θα πρέπει να θεωρηθεί ότι πρέπει να εξεταστεί. Εκεί όπου πρέπει να γίνει κάτι για να γεφυροποιηθούν αυτές οι διαφορές πρόσθετα κονδύλια απαιτούνται. Γι' αυτό με εκπλήσει κάπως ότι στο τέλος τέλος από ό,τι φαίνεται στην τεχνογνωσία υπάρχουν ελλείψεις αλλά όσον αφορά τις χώρες συνοχής θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουν αυτά τα κονδύλια να διασφαλιστούν. Αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα τα κονδύλια αυτά ή τουλάχιστον να διασφαλιστούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος αυτών των κεντροανατολικοευρωπαϊκών κρατών. Γι' αυτό ερώτησή μου, τι γίνεται με τα διασυνοριακά αυτά προγράμματα και σχέδια. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι κάνετε λόγο συχνά για το blending, συνδυασμό ή μείγμα επενδύσεων, κονδυλίων ποια είναι η ε, αναλογία και πώς πρέπει να προχωρήσουμε με τέτοιου είδους συνδυασμούς ε, ώστε με αυτή την ε, περίοδο όσον αφορά τις προσδοκίες από πλευράς του ΕΦΣΥ και του ΣΕΦ για τα δισεκατομμύρια που απαιτούνται πρέπει προσπάθειες να γίνουν. Επιπλέον κονδύλια πρέπει να μπορέσουν να διασφαλιστούν μπορεί κανείς ε, να βασιστεί στο ότι σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσουν να διατεθούν αυτά τα κονδύλια από το ΕΦΣΥ για τον μηχανισμό διασύνδεσης της Ευρώπης. Αυτή είναι η ερώτηση που θα ήθελα να σας θέσω. Ευχαριστώ. σε ευχαριστώ. Εσείς τώρα έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για την παρουσίαση και για τα καλά σα λόγια. Έχω μία ερώτηση σχετικά με την παρουσίαση και με το πρόγραμμα εργασίας. Ή στο ΕΦΣΥ. Θα έχουμε μία δέσμη περί τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Και εξ όσων γνωρίζουμε τώρα, 50 δισεκατομμύρια αναφέρονταν τον Ιανουάριο. Άρα μιλούμε για ένα μικρό κομμάτι του συνολικού προϋπολογισμού. Επομένως ο σύνδεσμος μεταξύ ΕΦΣΙ και του προγράμματος της διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη, το CF, είναι αντιληπτός. Αλλά πώς θα λειτουργήσει αυτό δημοσιονομικά, αν θέλετε, ή χρηματοδοτικά. Θα ήθελα να ακούσω μια εξήγηση από αυτού. Δηλαδή εγώ αυτά που είχα ακούσει είναι ότι ο ΕΦΣΙ δεν έχει επαρκή κονδύλια. Πώς επομένως θα δοθεί η στήριξη αυτή. Γιατί μάλλον δεν έχει γίνει τόσο καλά όσο θα, είχε, όσο θα επιθυμούσε ο πρόεδρος Γιούγκερ. Τώρα για τα σχολεία του κ. Βάντεκα πριν από λίγες εβδομάδες ε, συμμετείχα σε μια συνάντηση με φορείς ε, των επιχειρηματιών όπου συζητήθηκε η δέσμη των μεταφορών και υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια σχετικά με το πότε θα υποβληθεί τελικώ αυτή η πρόταση. Μήπω θα μπορούσατε να μα δώσετε πιο συγκεκριμένε πληροφορίε για την ημερομηνία τη ειδικά τη δέσμη για τα οδικά. Επίση, από 1η Απριλίου το Βέλγιο εισήγαγε ένα τέλος για τις μεταφορές εμπορευμάτων στο δικό δίκτυο και από ό,τι ξέρω πρόκειται να επιβληθούν ε, τέλη και για τους επιβάτες. Αυτό θα οδηγήσει σε μεγάλη σύγχυση. Και οι επιχειρηματίες χρειάζονται ε, σαφήνεια. Χρειάζονται ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή τέτοιων τελών ή άλλων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η Γκεζίνε είναι το παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και σας Επίτροπε για την έκθεσή σας. Όπως και ο κύριος Φαντάλεν, έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις ε, για το ΕΦΣΥ και για τις χρηματοδοτήσεις ε, που αναφέρατε στην παρουσίασή σας και το άλλο που αφορά το πρόγραμμα εργασίας 2016-2017 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Μεταφορές. Γενικά δηλαδή στις ε, επενδύσεις συμβαίνει ότι αν παρατηρήσαμε και το είπατε ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ζήτηση από τις ε, δυνατότητες που είχαμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Είναι κρίμα το ότι σχετικά λίγο με καινοτόμες επενδύσεις ε, ε, ασχοληθήκαμε. Project, project bonds δεν έχουν προαχθεί, δηλαδή ε, τέτοια ομόλογα έργου για παράδειγμα και πώς μπορεί να λειτουργήσει το χρήμα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Να υπάρχει μόχλευση για παράδειγμα, 20 πλάσια μόχλευση σε σχέση με τη διάθεση των κονδυλίων. Όταν έχουμε 6,7 δις ευρώ που χρησιμοποιήθηκαν και συγγνώμη, 12,77 δις, δηλαδή περίπου 13 δις λοιπόν, 13 δις και 28 όσον αφορά τις επενδύσεις, περίπου το διπλάσιο, αλλά δεν ανταποκρινόμαστε στο στόχο που είναι περίπου 20 πλάσιος. Πώς μπορεί να λειτουργήσει η ευφυής καινοτομία στις επενδύσεις για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να βελτιωθεί η κατάσταση. Αυτή είναι μια ερώτηση που θα ήθελα να απευθύνω όσον αφορά τα χρήματα οικονομικά. Παράλληλα με τον Ισμαήλ υπάρχει ένας κατάλογος πόσα από αυτά τα προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν που περίπου ήταν 230 όπως αναφέρθηκε τι γίνεται με τα διασυνοριακά θέματα, τα missing links, ε, τους ε, απόντες κρίκους ε, για παράδειγμα και για τα, τους σιδηροδρόμους. Έχω την εντύπωση ότι τα κράτη-μέλη ζητούν πολλές φορές πράγματα που αφορούν το εθνικό τους επίπεδο περισσότερο, το εθνικό επίπεδο κρατών μελών και όχι τόσο διασυνοριακά σχέδια και προγράμματα. Και για τα όσα παρουσιάζονται π.χ. για το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης και πρέπει να δούμε εδώ το θέμα της ε, διασυνοριακής συνιστώσας και να δούμε και τους ε, ε, κρίκους που απουσιάζουν σε αυτή τη διασύνδεση της Ευρώπης. Και Θέλω να ακούσω την άποψή σας. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούν να γίνουν υπό το ευρωπαϊκό πρίσμα. Υπάρχει λοιπόν ένας κατάλογος, ένας πίνακας προτάσεων που θα μπορούσε να απορρεύσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα έπρεπε εμεί ως Ευρωβουλευτές να κάνουμε σε σχέση με τις εθνικές κυβερνήσεις να ασκηθεί κάποια επιρροή σε σχέση με τη Γερμανία. Γνωρίζω αυτού του είδους τις δραστηριότητες, φτάνουν μέχρι τα σύνορα αυτές οι δραστηριότητες, αλλά μετά πρέπει να δούμε και τις διασυνοριακές ανάγκες. Δεν είναι μόνο ε, ενδιαφέρον και συμφέρον της Γερμανία, μόνο να υπάρχουν ε, cross-border links, να υπάρχουν διασυνοριακοί δεσμοί. Χρειάζονται αυτοί οι δεσμοί και αυτές οι διασυνδέσεις διασυνοριακά. Πώς μπορούν να αποτροχοπεδηθούν λοιπόν, να απελευθερωθούν αυτές οι δυνατότητες. Αυτό θα ήθελα να μου πείτε από πλευράς χρηματοδότησης και από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι συγκεκριμένα το ερώτημα για το 2017. Πότε θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε για το 2018 και να μπορέσουμε να δούμε και το ερώτημα τι γίνεται με το road package, τη δέσμη μέτρων για τις ε, οδικές μεταφορές. Ε, παράλληλα με τις άλλες δραστηριότητες, ε, αυτή η δέσμη μέτρων ε, όσον αφορά το, τις δραστηριότητες για τον τομέα των οδικών μεταφορών πρέπει όχι ε, ε, μεμονωμένα αλλά σαν ένα σύνολο να εξεταστούν και να δούμε και με ποια σειρά θα μπορέσουμε να δράσουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριε, παρακαλώ ευχαριστώ κυρία Κιλέναν. Ευχαριστώ κυρία Μπούς για την παρουσίαση, για τις ε, ερωτήσεις ε, που απορρέουν. Ερωτήσεις. Ε, είσαστε ικανοποιημένοι με την ποιότητα, το επίπεδο των κονδυλίων και των δράσεων και σε σχέση με τα όσα έχουν αναφερθεί για την ε, ε, εφαρμογή όλων αυτών και την, ε, τις πληροφορίες που έχετε ανταποκρίνεται το επίπεδο αυτό στις προσδοκίες σας όσον αφορά τις ανάγκες και πώς βλέπετε την συζήτηση που διαμορφώνεται όσον αφορά την αποανθρακοποίηση, την ε, ε, ελάφρυνση του περιβάλλοντος από τον άνθρακα για ιδέες που πραγματικά θα μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα να επιτύχουμε τον στόχο της μείωσης ε, του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ή επιλεκτικά συλλέγουμε κάποια στοιχεία ώστε να δράσουμε επιλεκτικά στο μέλλον πώς μπορούμε να όλες τις δυνατότητες και εναλλακτικέ λύσεις να τις κρατήσουμε ανοιχτές. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο μας απασχολεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και αυτό είναι πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το να ε, έχουμε πληροφορίες και στοιχεία για τα προγράμματα υποστήριξης και αρρωγής και πώς μπορεί να βελτιωθεί και ο συντονισμός αυτών των προγραμμάτων μεταξύ τους. Εμείς ως Ευρωβουλευτές φυσικά ε, μας ενδιαφέρει άμεσα το να έχουμε αυτές τις πληροφορίες ε, για να είμαστε αποτελεσματικοί αλλά ακόμα περισσότερα χρειάζονται στην επικοινωνία και στο συντονισμό μεταξύ των εμπλεκών και θα ήθελα σε σχέση με την ερώτηση που διατυπώθηκε να δούμε την δυνατότητα απάντησης. Πώς μπορεί να υπάρξει ένα ενωμένο μέτωπο, ένα ενωτικό μέτωπο για να μπορέσει να ε, βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά την αηφορία των μεταφορών και να είναι δυνατόν να προχωρήσουμε και με βάση τις προτάσεις και των Ολλανδών συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και την Επίτροπο που ήταν εδώ μαζί μας για να μας παρουσιάσει όλα αυτά τα στοιχεία για κάποια έργα. Βλέπω όμως εγώ αυτά τα έργα που είναι στο σχεδιασμό του Ταμείου για τα Στρατηγικά, από τα οποία έχουμε τρία για επεκτάσεις αυτοκινητοδρόμων, το οποίο το έλεγξα και στην ε, ιστοσελίδα της τράπεζας, γιατί εδώ έχουμε ένα πρόβλημα σε σχέση με τη Γαλλία. Από ό,τι βλέπουμε λοιπόν είναι ότι ούτε η τράπεζα ούτε και τα κράτη-μέλη δεν παίζουν το ίδιο παιχνίδι σχετικά με τη χρηματοδότηση τέτοιων έργων. Ωστόσο είχε δοθεί ένα πολύ σαφές πολιτικό μήνυμα προς την τράπεζα με συγκεκριμένους στόχους και αντικείμενα για επενδύσεις στρατηγικού επίπεδου σχετικά με τη μόνιμη κινητικότητα, τη χρήση νέων τεχνολογιών κτλ. Και επομένως διερωτώ με πώς μπορούμε να δεχθούμε ότι μετά τις συμφωνίες του Παρισιού για το περιβάλλον, για το κλίμα και υπό το φως της ανακοίνωσης της δικής σας για την απομάκρυνση από τον άνθρακα επενδύουμε ακόμα στην τεχνολογία των αυτοκινητοδρόμων το 2016. Γιατί τελικά είναι η δική μας γενεά, η δική μου γενεά που θα χρειαστεί να πολεμήσει για να συγκρατήσει την κλιματική αλλαγή. Πώς λοιπόν υπολογίζουμε ώστε θα υλοποιήσουμε αυτήν την εντολή που εδόθη προς την τράπεζα. Για να επανέλθω τώρα στα του μέλλοντος. Θα μπορούσατε, Επίτροπε, να μας επιβεβαιώσετε το τι τελικώς θα γίνει για την δέσμη των οδικών και μιλώ για δύο ε, διατάξεις. Την οδηγία σχετικά με το εξωτερικό κόστος και άμεσες, άμεσους σχετισμούς με την ε, περιβαλλοντική αλλαγή και επίσης θα είναι σημαντικό θα είναι σημαντική αυτή, δηλαδή θα ληφθεί υπόψη σε σημαντικό επίπεδο αυτή η οδηγία. Επίσης, σκοπεύεται να εντατικοποιηθεί η συγχρηματοδότηση των συνδέσμων των περιφερειακών και των κενών που έχουμε στις ε, συνδεδρομικές ενώσεις. Και επίσης οι επενδύσεις των υφισταμένων γραμμών θα συνεχίσουν ή όχι. Γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Τελικώς σήμερα έχουμε ένα όραμα, ένα προγραμματισμό, κάποιους στόχους σχετικά με κάποια κενά που έχουν σημειωθεί ή στην ασφάλεια κυρίως των αερολιμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα είναι τμήμα των σχεδιασμών σας και των στοχεύσεών σας για το υπόλοιπο του έτους. Ευχαριστώ κυρία Επιτροπή. Ευχαριστούμε. Πέτερ Λούντγκρεν τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση για διάφορα προγράμματα, αλλά ε, προσπαθούμε να καταλάβουμε όλοι τι θα κάνουμε στο μέλλον και πού θα βρούμε τα χρήματα τα οποία χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε συνεργασία με τις χώρες μας και ξέρουμε ότι Υπάρχουν ε, κολλήματα για διάφορες προτάσεις. Ε, μπορώ να σας πω όμως ότι έχουν βαρεθεί όλοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λένε «Α, πρέπει να επιτύχουμε εκείνο και το τάδε και το δίνα» αλλά έχουν βαρεθεί όλα ή διότι δεν αντιμετωπίζονται τα βασικά τους προβλήματα, τα καθημερινά τους προβλήματα. Παραδείγματο χάρη, καλέ, ε, τα προβλήματα που έχουμε και πέρα ε, χτυπιούνται, αγωνίζονται όλοι στη ζούγκλα του καλέ για να επιβιώσουν. Και εμεί τι κάνουμε, προσπαθούν να περάσουν στην Αγγλία. Για με τέτοια πρέπει να ασχολούμαστε ε, ε, και με αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να λύσουμε. Επίσης, στην Σουηδία για να έχουμε περισσότερους δικαιούχους. Ε, να μας πείτε τι θα κάνουμε με το παράνομο καμποτάζ. Ε, ε, βλέπουμε ότι εκατοντάδες ε, Σουηδοί ε, συμμετέχουν σε αυτό το λαθρεμπόριο, στο παράνομο καμποτάζ ε, και πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η λύση, να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι και με πυγμή να διεκδικήσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Χρειαζόμαστε δηλαδή αποφασιστικότητα από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρόλα, πα, αυτά τα προβλήματα περιοριζόμαστε σε ευχολόγια, σε οράματα. Αυτά τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και μάλιστα τώρα, όπως είπαν και διάφοροι άλλοι συνάδελφοι, χρειαζόμαστε επίση ε, πληροφορίε σε σχέση με τι οδικέ ε, μεταφορέ, ε, γιατί αυτό είναι διαφορετικό πακέτο και θα ήθελα λοιπόν, επειδή για μα είναι επίγον το πρόβλημα, να ακούσω αν υπάρχουν πρωτοβουλίε και συγκεκριμένε λεπτομέρειε για τι οδικέ μεταφορέ. Και πρώτα απ' όλα, όπω και άλλοι, θα ήθελα να ξέρω πότε ακριβώ θα υποβάλλεται συγκεκριμένο το πακέτο των οδικών μεταφορών, συγκεκριμένη πρόταση. Ευχαριστώ. Κριστίν Ρεβουνταλόν, παρακαλώ. Merci. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επίτροπο για την παρουσίασή τη. Ε, πρώτα απ' όλα, είχατε, αναφερθήκατε στο, στο Τιουχέλ που ήταν ένας πρώτος διαγωνισμός και ένα πρώτο βήμα που μας οδηγεί προς τα εμπρός. Αυτό είναι ικανοποιητικό. Τώρα για τα CEF είχαμε εκφράσει μια απογοήτευση για τη μείωση του 2015 και εξακολουθούμε να στηρίζουμε ότι θα επανέλθουμε στο προηγούμενο επίπεδο το επόμενο έτος ή στα πλαίσια της επόμενης αναθεώρησης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Τώρα για το ΕΦΣΥ. Η ερώτηση αυτή ετέθη ήδη από τους συναδέλφους κατά τον τρόπο αλλά ε, εγώ θα επιθυμούσα κάποιες περισσότερες απαντήσεις σχετικά με τα έργα που δεν είναι στο εσωτερικό δίκτυο, αλλά στα υπόλοιπα δίκτυα. Δηλαδή στα δίκτυα που έχουμε, δεν έχουμε τόσο ικανοποιητική προσβασιμότητα σήμερα. Προβλέπετε κάτι συγκεκριμένο ώστε και αυτά τα έργα να μπορέσουν να επιτύχουν μια στήριξη. Όσο δε για τα έργα στα οποία παρεμβαίνει απευθείας η τράπεζα, είδαμε στην παρουσίασή τη ότι έχουμε ένα σχετικά περιορισμένο αριθμό. Γιατί, ποιος είναι ο λόγος αυτού του περιορισμού. Ιδιαίτερα αν μιλούμε για έργα τα οποία στο παρελθόν λιγότερο είχαν συμμορφωθεί προς τους οδικούς χάρτες και τις συστάσεις της Κομισιόν. είχαν εξευρεθεί κάποιες ιδιωτικές επενδύσεις και γι' αυτό είχαν διευκολυνθεί. Αλλά μήπως έργα που είχαν συμμορφωθεί καλύτερα από τις διατάξεις τελικά έχουν αφαιθεί στο περιθώριο. Σας ευχαριστώ Ντομινίκ Ρικέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επίτροπο για την θαραλέα της επίσκεψη. Θαραλέα, πρέπει να το πούμε. Συμμερίζομαι και εγώ κάποια σχόλια των συναδέλφων για το πρόγραμμα εργασία και θα περιμένω και εγώ να ακούσω κάπως περισσότερα πράγματα και για τις δέσμες και τον περιεχόμενο τους. Έχουμε και κάποιες νομοθετικέ προτάσει κανονισμών και τα λοιπά και μια σειρά από στοιχεία. Και είναι αλήθεια ότι όλα τα είδη μεταφορών ενέχονται. για το πρόβλημα των επενδύσεων, το ζήτημα των επενδύσεων, που απασχολεί κάποιους από εμά ιδιαίτερα. Αρχίζουμε στα, στις μεταφορές να έχουμε κάποια αποτελέσματα ενδεχομένω από το σχέδιο Juncker και είχαμε δύο είδη επενδύσεων. Δηλαδή ένα επικερδές έργα ώστε να έχουμε και μια επιστροφή της επένδυσης. Αυτή είναι η βασική αρχή. και υπάρχουν αποδόσεις αν θέλετε και επιστροφές και άλλου είδους από το χρηματοδοτικό κοινωνική ε, ωφέλεια κτλ. Τώρα ε, μεταξύ αυτών υπάρχει ένα δημόσιο ενδιαφέρον ή συμφέρον επί της απόδοσης αλλά η απόδοση αυτή θα πρέπει τουλάχιστον να καλύπτει το κόστος του κεφαλαίου. Τουλάχιστον το κόστος του κεφαλαίου. Γιατί το κεφάλαιο κοστίζει και αυτό. Η παροχή του. Και υπ' αυτήν την έννοια τοποθετούμε, γιατί έτσι είχα καταλάβει ότι θα λειτουργούσε το σχέδιο του Γιούνκερ. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι επενδύσεις για τις οποίες έχουμε πρόσθετα στοιχεία. Δηλαδή, δεν είμαστε στην οικονομία της αγοράς και πρέπει να ενισχυθεί κάποιο στοιχείο ώστε να προσελκυθεί το ιδιωτικό κεφάλαιο. Αυτές οι διευκολύνσεις ή τροποποιήσεις είναι πολύ σημαντικές σε σχέση με στοιχεία που έχουν άμεσο δημόσιο συμφέρον. Από την άλλη όμως από όλα τα έργα που αναφέρθηκαν εδώ σήμερα ε, για ζώνες που δεν είναι συνδεδεμένες ε, είναι προφανές ότι δεν είναι επειδή δεν έχουν ε, οικονομικό ενδιαφέρον προσέλκυσης. Για διασυνοριακά ή ευρωπαϊκό επίπεδο, για τις διευκολύνσεις για περιβαλλοντικά στοιχεία όλα αυτά γιατί δεν γίνονται φυσικά, αν θέλετε, από μόνα τους. Γιατί δεν εμπίπτουν στην οικονομία της αγοράς. Αλλά το βασικό αμάρτημα του σχεδίου Γιούνκερ και το είχα ήδη πει αυτό, είναι ότι δεν μπορούμε μόνο στα στοιχεία προστατικότητος των χρηματοδοτικών μέσων να βασίζουμε τη στόχευσή μας. Δηλαδή, είχαμε ακούσει πολλά εφάνταστα στοιχεία, project bond, υποχρεώσεις, ενδιάμεσης, ε, equity, ή μη equity κτλ. Όλα αυτά όμως για να έχουμε επαρκή αποτελεσματικότητα δεν επαρκούν. Χρειάζονται ενισχύσεις και πέρα της περιβαλλοντικής διάστασής τους ή της καθαρά χρηματοπιστωτικής τους διάστασης. Άρα, όταν φτιάξαμε τον ΕΦΣΥ, τι κάναμε. Πήγαμε να βρούμε κονδύλια εκεί που υπήρχε διαθεσιμότητα ενισχύσεων και αν θέλετε καπιταλιστικού ενδιαφέροντος. Αυτά όμως τα προσθέσαμε σε έργα που δεν θα είχαν κυλήσει φυσικά από μόνα τους και χωρίς βοήθεια. Και αν κοιτάξουμε τα έργα του ΕΦΣΙ δεν θα βρούμε στοιχεία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Δεν θα βρούμε στοιχεία δημοσίου συμφέροντος και ε, παρατηρώ, σημειώνω, ε, το γράφημα αυτό που έχετε φτιάξει εδώ, το διάγραμμα, έχει μια ενδιαφέρουσα ε, προβολή φαντασίας. Λάβαμε το 30% της δυνατότητας επενδύσεων για την Connecting Europe Facility, 30% για τις μεταφορές, εντός του οποίου υπάρχει 5% πρόσθετα στοιχεία, προσθετικότητες προστεδεμένα στοιχεία, για τα οποία όμως δεν επαρκεί αγορά, δεν θα λειτουργήσει. Χρειάζονται ενισχύσεις. Αναφερθήκατε στο λιμάνι του Καλέ, που το γνωρίζω καλά. Το έχω εργαστεί για χρόνια. Υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ εντός του ΕΦΣΥ, αλλά επειδή υπάρχουν, υπάρχει υψηλό επίπεδο ενισχύσεων που καθιστούν, αν θέλετε, την υλοποίηση του έργου δυνατή. Και σχετικά με το Ρότερνταμ, εγώ θυμάμαι το 2009 είχα συμμετάσχει στη συνάντηση της Ραγώσας και είχα προτείνει τότε να δημιουργήσουμε ένα ταμείο ενισχύσεων για να προσελκύσουμε τις επενδύσεις. Που τότε μιλούσαμε για 80 δισεκατομμύρια και τότε με κοιτούσαν σαν να είχα έρθει από τον Άρη οι συνάδελφοι. Και στο CEF όταν είδαμε τα, τα, τα, ποσά, τα κονδύλια να περιορίζονται ακόμα περισσότερο μετά τις μεταφορές που έγιναν, το ερώτημα που τίθεται είναι φαντάζομαι ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε 300 δις ε, επενδύσεις λόγω των αναγκών που υπάρχουν. Θα καταφέρουμε και κάποια συνδεδεμένα στοιχεία. Αλλά μιλήσαμε για 30%, 30% για τις μεταφορές. εδώ είμαστε στα επίπεδα του 15. Και μόνος επίτροπε φοβούμε τελικώς εάν συνυπολογίσουμε τις, ε, τα προσδεδεμένα στοιχεία θα καταλήξουμε σε κάτω του 10%. Κάτω του 10%. Διότι αν αφαιρέσετε τις ενισχύσεις αφαιρείτε την ρεαλιστική υλοποιησιμότητα των έργων αυτών, των επενδύσεων αυτών. Η Τράπεζα Επενδύσεων προχώρησε σε μια ε, χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική των έργων αυτών, των προγραμμάτων αυτών. Εδώ μιλούμε για χρηματοδοτήσεις δημοσίου ενδιαφέροντος, στοιχεία δηλαδή που δεν λειτουργούν πάνω από μόνα τους στην αγορά την καπιταλιστική, στην ε, οικονομία της αγοράς, Επομένως δεν έχουμε βασίσει την όλη δομή σε αυτά που μας ενδιαφέρουν εμάς και στις μεταφορές. Ευχαριστώ. Μάκους Πίπα. Μάκους Πίπα. Ευχαριστώ Επίτροπε. Θα ήθελα και εγώ ε, να σχολιάσω ε, κάποια θέματα σε σχέση ε, με αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι. Ας δούμε τι έγινε την ε, τελευταία 15 ετία. Υπέροχα προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν με ευρωπαϊκές επιδοτήσεις ε, και αυτά, αυτοί ήταν οι στόχοι τους, εκπληρώθηκαν. Είναι καταπληκτικά αυτά που έχουμε καταφέρει την τελευταία 15 ετία. φυσικά έχουμε Ε, αυτή την υπερηφάνεια, ε, για αυτά που έχουμε καταφέρει, όμως ξεχνάμε ενδεχομένως το στόχο το βασικό μας στόχο για τα σιδηροδρομικά δίκτυα, για τις ε, οδούς, εσωτερικές πλωτές οδούς και ε, Επίση, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν ε, έχουμε τρία διαφορετικά προγράμματα για αυτοκινητοδρόμου, ούτω ή άλλω θα είχαμε βρει ιδιωτική χρηματοδότηση, ακόμη και αν δεν καλύπτονταν από το ΕΤΣΕ. Τι γίνεται λοιπόν με αυτά τα προγράμματα. Έχουμε τα προγράμματα που καλύπτουν τα λιμάνια. Αναφερθήκατε στο καλέ. Είναι πολύ σημαντικό για του ε, ιδιώτε επενδύτε, διότι υπάρχει εγγύηση από το γαλλικό κράτο Οπότε λυπάμαι, όμως ε, θεωρώ ότι βασιζόμαστε σε ε, προγράμματα που... Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει, να διασφαλιστεί η πρόσθετη χρηματοδότηση, αλλιώς δεν γίνεται. Από την Επίτροπο για τις Μεταφορές θα ανέμενα ότι θα ενδιαφερόταν περισσότερο για αυτούς τους τομείς και θα έλεγε ότι αυτά που έγιναν με το ΣΕΦ, αυτά που συνέβησαν με το ΣΕΦ δεν έβαιναν καλώς. Και εγώ ως Επίτροπος θα καταβάλω κάθε προσπάθεια ώστε αυτός ο τομέας να καλυφθεί, να πληρωθεί και καλυφθεί όπως πρέπει και να επεκταθεί στην νέα κοινοβουλευτική ε, περίοδο όπως πρέπει. Αυτό θα ανέμενα από την αρμόδια Επίτροπο. Μια και γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ε, δημοσιονομικές διαπραγματεύσεις 2016 δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματική. Δεν είναι πλάκη όπως έπρεπε. Δεν ξέρω ποιος είναι εκείνος ο οποίος ισχυρίστηκε ότι τα χρήματα για το σέφα δεν θα χρειαζόντουσαν λέει επιπλέον. Και ε, υπήρξε και επιστολή σε σχέση με τον Πρόεδρο για αυτό το θέμα αναφέρατε ότι υπάρχει λέει τριπλάσιο σε σχέση με, το, με τη ζήτηση. Πώς μπορείτε να ισχυριστείτε κάτι τέτοιο ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα έπρεπε να, να είχατε περισσότερο θάρρος ως Επίτροπος για τα θέματα μεταφορών και να καταβάλλετε προσπάθειες ώστε αυτά τα θέματα να διασφαλιστούν. Στρεφόμενοι προς τα επόμενα έτη, προς το μέλλον και τις ε, δημοσιονομικές διαπραγματεύσεις πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις πλωτές μεταφορές, με τα συνδρομικά δίκτυα, με τις οδικές μεταφορές όταν ε, υπάρχουν ίσως κάποια ενδιαφέροντα και συμφέροντα κάποιων επενδυτών. Πρέπει όμως εδώ να δράσουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Μαρή Κριστίνα Ροντή, παρακαλώ. Merci, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Ε, Σα ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Ε, κάποιε παρατηρήσει. Ε, αυτή η ιδέα του κυρίου Γιούγκερ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, όπω είπαν και οι συνάδελφοι, αυτή καθ' αυτή δεν ήταν κακή. όμω αν κρίνουμε από τα πρώτα αποτελέσματα, μπορεί κάποιο να θεωρήσει ότι μάλλον για αποτυχία πρόκειται. Διότι με πολύ δυσκολία καταφέρει να τονώσει την οικονομία των κρατών μελών και να πείσει του ιδιώτε επενδυτέ ε, αποδείξει για να μείνω στον τομέα των μεταφορών, η χρηματοδότηση τη γραμμή γραμμή σε το Ρήνο. Ε, ε, ζητάνε χρήματα από το Έτσε, από τον Γιούνκερ, ε, από πλευρά Ιταλία και η Γαλλία τα αντιλεί από το ΣΕΦ. Και το ΣΕΦ έχει χάσει πολλά κονδύλια λόγω του Γιούνκερ, δηλαδή η γάτα που δαγκώνει την ουρά τη α πούμε. Θα πρέπει να δούμε επίσης ότι πολλά έχουμε υπερβεί τις προβλέψεις μας για τα προγράμματα ή δεν έχουν επαρκή ευρωπαϊκή διάσταση είναι τόσο ισχνή που τελικά καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ε, και πάλι περιτεύει η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση γιατί τα κράτη και η ΟΤΑ θα είχαν ούτως ή άλλως μέσα για να δράσουν για τους αυτοκινητοδρόμους παραδείγματος χάρη. Είναι σουρεάλ να διαπιστώνουμε ότι ε, χρηματοδοτούνται ακόμη προγράμματα οδικών μεταφορών. Ε, για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίρνει χρήματα από το ΣΕΦΕ για προγράμματα που σχετίζονται ε, με το μετρό στο Παρίσι ή στη Λιόν, παραδείγματο χάρη. Ε, και το ίδιο έτσι το έτσι μάλλον ε, αντικαθιστά ε, δημόσια ε, χρηματοδότηση που ήδη προβλέπεται, παραδείγματο χάρη στη Γαλλία για το, το δυτικό Στρασβούργο προβλέπεται παράκαμψη, δεν δημιουργεί πολλές θέσεις απασχόλησης και εντάξει νόνι το διασυνοριακό εμπόριο και από ό,τι φαίνεται αυτός είναι ο μοναδικός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν βλέπουμε κανένα ενδιαφέρον. Επίσης να πούμε για τη Γαλλία που είναι ο δεύτερη στη σειρά ω ε, τη συνεισφορά στον προπολογισμό. βλέπουμε ότι εποφελούμαστε με ένα από τα κονδύλια όμω θα πρέπει να τηρείται και η αρχή τη επικουρικότητα, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτού ε, του ε, θάλαμου αερίων όπω λέμε και τελικά αυτή τη μαύρη τρύπα όπου χάνονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, έχω εγγράψει τον εαυτό μου στον κατάλογο. Α, εσείς όμως πρώτα, παρακαλώ. Eh, er Ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομο πράγματι, επειδή πολλά ερωτήματα ήδη διατυπώθηκαν. Και θέλετε κι εσείς ε, να παρέμβετε. Λοιπόν, να υπάρξει και αρκετός χρόνος να απαντήσει και η Επίτροπος. Το εξής, η προσέγγιση που θα υιοθετηθεί σε όλα αυτά τα προγράμματα και σχέδια υπό το ΕΦΣΥ τι νομίζετε σε σχέση με την ε, ε, επικέντρωση και μετάθεση ε, επικέντρωσης, τι μπορεί να γίνει. Υπάρχουν όμως πολλά προγράμματα για τις οδικές μεταφορές που αναφύονται και ο πολλαπλασιαστής είναι χαμηλότερος και όταν βλέπουμε από 1 έως 15 πολλαπλασιαστές και βλέπουμε ότι σήμερα υπάρχουν πολλαπλασιαστές 1, προς 2, 1 προς 3 τι γίνεται όμως με την ποιότητα αυτών των προγραμμάτων σε σχέση με τα όσα έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα χωρίς ε, τα κονδύλια του ΕΦΣΥ και τι θεωρείται σε σχέση με τους πολλαπλασιαστές ε, για τη μόχλευση. Είναι πολύ χαμηλός ο, ε, η επίπτωση του πολλαπλασιαστή σε αυτά τα επίπεδα είναι πολύ χαμηλή. Δεν θα πρέπει να αναζητηθούν άλλες δυνατότητες. Ευχαριστώ. Yeah, Πρόεδρος, ευχαριστώ. Τώρα έχω εγγράψει εγώ τον εαυτό μου στο τέλος τέλος και πρόκειται όχι μόνο για χρήματα φυσικά εδώ, αλλά με το πρόγραμμα Juncker τρεις στόχοι ακολουθούν. Πρώτον, η καταπολέμηση της ανεργίας. Θέλαμε με στοχοθετημένα σχέδια να αναχαιτήσουμε τις κλιματικές αλλαγές και θέλαμε να ολοκληρώσουμε την ευρωπαϊκή διάσταση. Το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης δεν έχει καμιά σχέση με ευρωπαϊκή συνιστόσα. Είναι καθαρά εθνική υπόθεση. Πώς μπορούμε λοιπόν με αυτά τα κονδύλια στοχοθετημένα να επενδύσουμε για την Ευρώπη. Εγώ προέρχομαι το Βερολίνο. Είχαμε πολλές κακές εμπειρίες όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου η απόφαση σε 30 χρόνια 5 χιλιόμετρα να δημιουργηθεί και όταν είχαμε τη δημιουργία του ε, τραμ ενώ ήταν χωρισμένη, διχοτομημένη η πόλη και μετά βλέπουμε σε σχέση με Θεσσαλονίκη κονδύλια σε ένα εγχείρημα για τη δημιουργία του μετρό έχουν διοχετευθεί που δεν προχωρούν όμως, δεν προχωρά αυτό το πρόγραμμα. Πώς μπορούμε γρήγορα, ταχαίως να δράσουμε ώστε να ολοκληρώνονται τα έργα και όχι να ε, λιμνάζουν. Ξέρουμε ότι εμβαλωματικά δρούμε στην Ευρώπη και σε σχέση με τα κενά που υπάρχουν χρειάζονται πιο στοχοθετημένες δράσεις. Πρότασή μου, σε σχέση με, το, ε, με τα σύνορα ε, και τη διασυνοριακή συνιστόσα να μπορέσουμε να δράσουμε με 85%. Πολλές χώρες θα έλεγαν εντάξει, ίσως αυτό δεν είναι πολύ, πιο, πολύ σημαντικό για μένα, αλλά εφόσον υπάρχουν χρήματα για τη διασυνοριακή διασύνδεση θα συμμετάσχω κι εγώ. Ή γνωρίζουμε όλα αυτά τα παραδείγματα όλοι. Αν επί 20 χρόνια στέλνουμε ε, γεωτρύπανα να διατρήσουν τα βουνά, τα όρη των Άλπαιων, ε, πρέπει να δούμε εδώ ότι είναι ένας κύριος λόγος για το πρόγραμμα Juncker να μπορέσουν να συγκεντρωθούν κονδύλια ώστε η ανεργία, κυρίως η ανεργία των νέων σε υψηλότατα επίπεδα να καταπολεμηθεί. Με αυτά τα προγράμματα λοιπόν να μην στρεφόμαστε μόνο στα κονδύλια, πιο ύψος κονδυλίων διατίθενται, αλλά να δούμε τι γίνεται με το κλίμα, ποιες επιπτώσεις υπάρχουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και υπάρχουν τεράστιες διαφορές λοιπόν αν συγκρίνει κανείς τέτοιου είδους ε, προγράμματα. Λοιπόν, αν δούμε σε σχέση για παράδειγμα με τις χώρες συνοχής ε, το ότι δεν υπάρχει ούτε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Είναι θλιβερή αυτή η κατάσταση. Όταν υπάρχει ένας freight corridor, ένας διάδρομος ε, φορτίων που από την Βαλτική θάλασσα ξεκινά και περνά μέχρι την ε, Μεσόγειο και μόνο μέσα από νέα κράτη-μέλη ε, περνά αυτός ο διάδρομος. Γίνονται προσπάθειες και από, κράτη, από παλαιότερα κράτη-μέλη να ε, υπάρξει παρέμβαση. Πόσο, πώς μπορεί να προχωρήσει αυτό. Γιατί δεν χρειάζονται εδώ σύραγγες, αλλά πρέπει να υπάρξει σε κάποιες διαδρομές μια δεύτερη σιδηροτροχιά ηλεκτροδότησή της ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πώς μπορείτε να υποστηρίξετε λοιπόν τέτοιου είδους δράσεις και όχι ε, τον 27ο ε, αυτοκινητόδρομο στη Γερμανία ή στη Γαλλία ή αλλού. Διασυνοριακή συνιστόση είναι πολύ σημαντική. Και τελευταίο σημείο, το πρόγραμμα εργασίας ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πλοία στις πρωτες μεταφορές χρειαζόμαστε τις την τεχνολογία ακόμα και όταν αντικατασταθεί, ακόμα και αν υποκαταστήσουμε το αργό πετρέλαιο από το ντίζελ πρέπει να δούμε τη διαφορά που θα υπάρξει. Εδώ θα υπάρξει πρόσθετο κόστος ίσως διότι όταν έχουμε το αργό πετρέλαιο, το βαρύ πετρέλαιο και αν υποκατασταθεί αυτό με, το ντίζελ θα είναι μια τεράστια πρόοδος. Δεν χρειάζονται τόσο, τόσο μεγάλα κονδύλια, θα είναι ίσως ε, μεγαλύτερα τα κόμιστρα υψηλότερα τα κόμιστρα για τη μεταφορά αγαθών με το ντίζελ. Αλλά μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τελευταίο, τελευταία παρατήρηση. Στην Σύνοδο των Προέδρων επανειλημμένα ασκήθηκε επίκριση στον κύριο Γιούνκερ και στον κύριο Τίμερμαν ότι δεν διαδραματίζει ρόλο το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ για την κινητικότητα και τα θέματα του κλίματος πρέπει να δράσουμε και πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Κάθε φορά θα το επαναλαμβάνω. Ερώτησή μου, πότε θα κατανοήσει εκεί πάνω η ψηλά ιστάμενη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι παλαιοί επίτροποι δεν έχουν τέτοια εμπλοκή όπως κατ' παρελθόν. Ποιο είναι το επιχείρημα εναντίον ώστε να μην διαδραματίζει ρόλο το θέμα των μεταφορών και να δούμε και το θέμα του περιβάλλοντος που έχει η θέμα ε, ρόλο επιβίωσης για μας να αναχαιτιστούν οι κλιματικές αλλαγές. Χρειάζεται όμως μια διαφορετική κινητικότητα και εδώ πρέπει να δράσουμε τα καταφέραμε σχεδόν, ε, τώρα μπορείτε να απαντήσετε στο χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας και προσδοκούμε να ακούσουμε τις απαντήσεις σας όλοι. Okay, first of all... Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους για όλα αυτά τα ποικίλα ζητήματα και παρατηρήσεις που έγιναν. Το οποίο μας αποδεικνύει για μία ακόμα φορά πόσο περίπλοκα και πολυδιάστατα είναι όλα αυτά τα ζητήματα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα μεταφορών σήμερα. Αυτό διατηρήστε το υπόψη. Ακόμα και τα δικά σας σχόλια μεταξύ τους αποκλίνουν. Πρέπει να βρούμε λοιπόν συνολικές λύσεις για την Ευρώπη. Αυτό δεν είναι εύκολο. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και νομίζω ότι βρισκόμαστε στην κατάλληλη κατεύθυνση. Τα έχουμε καταφέρει όλα. Όχι. Αναπτύσσουμε νέα εργαλεία, νέα μέσα. Ανοιχνεύουμε τα προβλήματα. Η έλλειψη του ανταγωνισμού είναι απολύτως προφανής στα συστήματα μεταφορών. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να έχουμε συστημική εικόνα, άποψη, να βλέπουμε τα κενά που υπάρχουν και που πρέπει να πληρωθούν ώστε να δημιουργήσουμε ένα καλά συνδεδεμένο σύστημα περιοχή μεταφορών που να εξυπηρετεί καλά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Σας άκουσα λοιπόν πολύ προσεκτικά. Εμείς σημειώνουμε και ενσωματώνουμε τις παρατηρήσεις σας προκειμένου να έχουμε αυτές τις συστημικές και βιώσιμες λύσεις που χρειάζονται. Είναι απολύτως σαφέ ότι υπάρχει και παραπληροφόρηση που κυκλοφορεί. Και πρέπει να δούμε πώς θα την περιορίσουμε. Γιατί σήμερα είναι δημοφιλές να λέει κανείς ότι δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές λύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να βρει λύσεις. Αν όμω μιλήσει κανεί με τους πολίτες απευθεία, όπως έκανα στη τελευταία μου επίσκεψη στην Πολωνία, ο κάθε ένα πολίτης από μόνο του, ασάρτητα, παραδέχεται ότι με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκή Ένωσης έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδο στη χώρα αυτή, που δεν θα μπορούσε να έχει γίνει εκτός της Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι αλήθεια για κάθε ένα από τα κράτη-μέλη. Όλοι έχουμε αποφεληθεί από την κοινή αγορά, από τους διάφορους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που έχουν δημιουργηθεί. Βεβαίως, δεν έχουμε κάνει όλα αυτά που θα επιθυμούσαμε και υπάρχει μελλοντική δυνατότητα ανάπτυξης. Αλλά 508 εκατομμύρια πολίτες είναι 508 εκατομμύρια πολίτες. Καμία χώρα από μόνη δεν έχει τέτοια δύναμη. 33 προϋπολογισμού καμία χώρα από μόνη της. Η δύναμη λοιπόν αυτή είναι της συλλογικής δράσης, της αποκοινού δράσης και πρέπει να διαμορφώσουμε τις συνθήκες ώστε οι μεταφορές να βοηθούν σε αυτήν την ανάπτυξη, σε αυτή τη μεγέθυνση, στη δημιουργία επιχειρήσεων που να είναι ανταγωνιστικές παγκόσμια και που να εξασφαλίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι και στο μέλλον όπως είναι σήμερα το καλύτερο σημείο διαβίωσης στον πλανήτη Γη. Να είναι και το μέλλον, γιατί σήμερα είναι. Δεν έχουμε βρει κάτι καλύτερο, λέει η Επίτροπος. Πρέπει λοιπόν να βρούμε νέους μηχανισμούς που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο. Ο καθένας από μας μπορεί να βρει μονομένες αφηγήσει που οδηγούν σε κενά, που διαπιστώνουν κενά, που οδηγούν σε δυσαρέσκεια, σε πρακτικές που δεν είναι δίκαιες, σε επενδύσεις που δεν έχουν γίνει με βάση τα καλύτερα δυνατά κριτήρια και γι' αυτό στο μηχανισμό CEF χρησιμοποιούμε πρότυπα της καλύτερης δυνατής διαχείρισης στο εσωτερικό της Κομισιόν. Έχουμε μια πολύ επαγγελματική επιλογή των έργων, πολύ επαγγελματική δομή διακυβέρνηση των προγραμμάτων αυτών. Και ναι, θα βελτιώσουμε τα πράγματα περαιτέρω, αλλά δεν γίνονται όλα σε μια, μια νύχτα, λέει ο Επίτροπο. Και βεβαίω πρέπει να συνεχίσετε με την επίκρισή σα. Μην μα αφήνετε στην ησυχία μα, αλλά στα βλέπουμε τα πράγματα επικοδομητικά και θετικά. Υπάρχει πάρα πολύ διακεχημένο αντιευρωπαϊκό πνεύμα αυτή τη στιγμή. Και αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα αποφεύγουμε. Εγώ, εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Εσάς σας αρέσουν αυτές οι τάσεις. Τουλάχιστον επ' αυτού ελπίζω να συμφωνούμε. Δηλαδή ναι κριτική. Ναι. Αλλά επικοδομητική. Ώστε να βρούμε λύσεις. Που θα μας κάνουν πιο δυνατούς και όχι το αντίστροφο. Τώρα στρέφομαι θα πάω και συγκεκριμένε ερωτήσει, αλλά ξέρετε συχνά είναι εκνευριστικό να προσπαθεί κανείς να βρει τις καλύτερες λύσεις και να αντιμάχεται διαρκώς αυτού του είδους τον γενικευμένο σκεπτικισμό που δημιουργεί σε απώλεια αν θέλετε ενέργειας, ε, όθησης για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε καλά. Λοιπόν, πολλές ερωτήσεις έγιναν για το πρόγραμμα εργασίας. Θα ξεκινήσω από αυτό γιατί μαζί με την απάντηση αυτή θα μπορούσα να απαντήσω και σε κάποια άλλα ερωτήματα. Πρώτον, λόγω της στήριξής σας έχουμε τη δύναμη αυτή τη στιγμή να ξεκαθαρίσουμε τον εκρεμή κατάλογο. Τον κατάλογο των εκκρεμών νομοθετημάτων. Η, η, η τέταρτη δέσμη δυναμικών. Πολύ καλή δουλειά έγινε εκεί, παρά τις, την κριτική. Έχουμε ένα φιλελεύθερο πλαίσιο για πρώτη φορά που επιτρέπει διευκόλυνση των προτύπων. 11.000 τοπικά πρότυπα αντικαταστάθηκαν από λιγότερο από 300 ευρωπαϊκά. Φανταστείτε πόσο αυτό θα διευκολύνει την ομαλή ροή των μεταφορών. Και ο πυλώνες αγοράς εισήχθη για πρώτη φορά για την εισαγωγή ανταγωνισμού και προσθέμενης αξίας υπηρεσίες. Δεύτερον, έμισα μια ανάπτυξη δυναμικού Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή, το οποίο προχωρεί και ελπίζω να έχουμε ολοκληρώσει σε λίγες εβδομάδε. υπηρεσίε λιμένων. Τον Ιούνιο ελπίζουμε ότι θα ολοκληρώσουμε το φάκελο αυτό για να προχωρήσουμε υπό μετά την Ολλανδική Προεδρία. Βεβαίω έχουμε για τα αεροπορικά και τα σλότ και διάφορα προβλήματα και καθυστερήσει. Δεν ξέρω πόσε φορέ μπορώ να το επαναλάβω, αλλά εμείς είχαμε επενδύσει στο ΣΕΖΑΡ για να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί συνολικά. Τώρα ο ανταγωνισμός χρησιμοποιεί πιο γρήγορα τα μέσα από ότι εμείς. Και ελπίζω πραγματικά ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα βοηθήσουν για να επιτρέψουμε στο οικοσύστημα των αερομεταφορών μας να προχωρήσει και να παραμείνει ανταγωνιστικό. Εν αυτό εκκρεμεί, δεν έχω καλά νέα από αυτού, δυστυχώς κοινά παραδοτέα για τις δεσμεύσεις του 16. Αναφερθήκατε πολύ συχνά στη δέσμη των οδικών, του δικού δικτύου. Εκεί προχωρούμε όπως είχαμε προσχεδιάσει. Είχαμε κάποιες εμπειρίες από πλευράς κομισιών και διοικητική δυνατότητα να προχωρήσουμε σε κάποιους φακέλους, αλλά χρειαζόμαστε τη δέσμη των οδικών γιατί. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να, μείνει, να παραμείνει ηγέτη στα αυτοματοποιημένα οχήματα και χρειαζόμαστε τη δέσμη αυτή για να εγκαταστήσουμε ευρωπαϊκές λύσεις που θα υποστηρίζουν αυτήν την νοοτροπία. Εδώ πρέπει να παραδεχθώ ότι παρότι έχω τοποθετηθεί πολύ συχνά στο θέμα αυτό, πολύ συχνά εγώ προσωπικά, μπορεί να έχουμε καθυστέρηση δύο μηνών, ας πούμε, σχετικά με την επιβεβαίωση του 8 συν 2 ίσως Φεβρουάριο-Μάρτιο. Αλλά σας παρακαλώ να βοηθήσετε κι εσείς, να πιέσουμε κι άλλο την Κομισιόν. Γιατί θέλουμε φέτος να έχουμε τελειώσει και να μην πάμε στο 17. Μιλούμε για ψηφιοποίηση. Η ηλεκτρονικά διόδια, ε, διασυνορικές υπηρεσίες, για πρώτη φορά εισαγωγή τέτοιων υπηρεσιών. Μιλούμε για το άνοιγμα της αγοράς, μιλούμε για κοινωνικά ζητήματα, με όλες τις προκλήσεις που υπάρχουν επιτάπτως εδώ, σε αυτό δηλαδή. Και άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες. Ιούνιος, η ασφάλεια των ε, σκαφών επιβατών. και μετά το CTIS Master Plan και στα τέλη του έτους νομοθετική πρόταση για την οδική ασφάλεια και για τα δικαιώματα των επιβατών για τις οδικές μεταφορές, για τις μεταφορές, συγγνώμη. Επίσης υπάρχει το fitness check, ο έλεγχος ε, που θα γίνει σε ενδιάμεσο στάδιο. Επίσης έχουμε στη συνέχεια τα προγράμματα για το μέχρι το 2017. Πρώτα απ' όλα ε, θα ε, ρίξουμε το βάρος το 2017 στις θαλάσσιες μεταφορές. Από συστημική σε πλευρά θα πρέπει να εξατεστεί η προσέγγιση μας αν να δούμε αν χρειάζεται κάτι περισσότερο ή θα, θα πρέπει να ε, προσφέρουμε κίνητρα για καλύτερη εφαρμογή. Θαλάσσιες μεταφορές αυτό θα είναι το κέντρο εστίας για το 2017. Για το 2018 και το 2019 θα είναι η πολυτροπικότητα, για να το ξέρετε. Ε, φτιάχνουμε την αρχιτεκτονική σε επίπεδο δεδομένων για την πολυτροπικότητα για να καταλάβουμε ακριβώς ε, ποια είναι τα κενά μας ούτως ώστε να συνδυαστούν όλοι οι τρόποι μεταφορών και για να έχουμε ολοκληρωμένη εφοδιαστική, ολοκληρωμένο σύστημα έκδοση εισιτηρίων και το καθεξής. Επανέρχομαι στα λάσια μεταφορές, ενδεχομένως του χρόνου θα μπορούσαμε να να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα και ξέρουμε ότι σε λίγες εβδομάδες, ίσως και μήνες, επειδή τώρα κάνουμε πέντε τέτοιους ελέγχους ε, fitness, ε, και το 16 ενδεχομένω να καταλήξουμε ή όχι σε νέε νομοθετικέ προτάσει σε υγεία, ασφάλεια, ψηφιοποίηση με απλούστευση των διατυπώσεων για την υποβολή αναφορών και μονοπευθυντική θηρίδα. Το είναι το βασικό, ε, το βασικότερο στοιχείο, δηλαδή χρειαζόμαστε μια σημεία επαφής ε, για τις θαλάσσιες μεταφορές ε, και επίσης υποδομές για τα για τα υπερπλοία, mega ships. και Άλλες σημαντικές ε, νομοθετικές ε, πρωτοβουλίες ε, για την μείωση των εκπομπών διοξιδίου, συνδυασμένες μεταφορές οδικές και σιδηροδρομικές και άρα συνδυασμός των διαδρόμων τους. να αναφέρω επίσης το ότι αξιολογούμε τώρα στα πλαίσια της συνεργατικής ε, οικονομίας, γιατί έπεται και η ανακοίνωση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χρειαζόμαστε νομοθετική πρωτοβουλία ε, για την πρόσβαση στα ταξί, στην αγορά των ταξί. Και το, θα ολοκληρωθεί η προσπάθεια μας το καλοκαίρι και θα εξετάσουμε αν χρειάζεται άνοιγμα της αγοράς για τα ταξί ή αν χρειάζεται να παρέμβουμε. Um, Ταυτόχρονα Υπάρχουν και μη νομοθετικέ δραστηριότητε, που είναι εξίσου σημαντικέ για το 2017. Σωστή εφαρμογή των εφισταμένων κανόνων, ε, νέοι δημοσιονομικοί κανόνε. Ε, θα λειτουργήσουν αυτές τις δραστηριότητες υποστηρικτικά για τους, ε, την υλοποίηση των στόχων μας. Αυτά. Ε, έκανα μια γενική επισκόπηση και ε, με μεγάλη χαρά να σας υποβάλουμε και γραπτώς απαντήσεις, τόσο ώστε όπως και σας προτείνατε να έχετε τα στοιχεία στη διάθεσή σας. Επόμενο σημείο και κοιτάζω και το χρόνο. Θα ήθελα, πέρα από την παρουσίαση αυτών των προγραμμάτων, να ε, απαντήσω σε κάποιες άλλες ερωτήσεις. Εύση. Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατηγικών Επενδύσεων έγιναν πάρα πολλά σχόλια και συμμερίζομαι τις ανησυχίες. Οφείλω να το πω και το εννοώ. Όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε μόνο μέσα από επιδοτήσει ανάγκες που έχουμε στον τομέα των μεταφορών. Τελεία. Και γι' αυτό προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Πρώτη φορά με το σχέδιο Γιούγκερ, πρώτη φορά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κινητοποιούμε ε, θεσμικούς επενδυτές. Φυσικά δεν τα κάνουμε όλα σωστά. Φυσικά κάνουμε λάθη, κάνουμε ε, ε, άσκοπες κινήσεις, το δρομούμε γιατί ξέρετε είναι μεγάλες οι δυσκολίες ε, διότι μιλάμε για εκατοντάδες ε, ε, προγράμματα και για το τέντι για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στο μέτρο μεταφορών πιστεύουμε ότι θα προωθήσουμε 50 τουλάχιστον προγράμματα. Είναι άλμα αυτό προς τα μπροστά και φυσικά έχουμε και πολλά οδικά προγράμματα. Αυτή ήταν όμως τα καλύτερα προετοιμασμένα και στο έτσι δεν έχουμε ακριβώς τους ίδιους κανόνες όπως για το ΣΕΦ για το Συνέδριο στην Ευρώπη. Καλά μου τα λέτε ότι χρειαζόμαστε τα, τα, χρήματα από το ΣΕΦ για το blending και άρα να εφαρμόσουμε και τους κανόνες του ΣΕΦ. Ναι, αλλά από την άλλη θα πρέπει να αποδείξουμε ότι λειτουργεί αυτό και ζητώ συγγνώμη, ήταν έτοιμα τα οδικά προγράμματα. Ίσως επειδή διότι μέσα από το ΣΕΦ δεν είχαν προηγουμένω δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν συγγνώμη, και το ΣΕΦ ε, είχε μάλλον κατευθυνθεί προς τι Μεταφορέ μεταφορές μέχρι στιγμής και έχουμε και τα διασυνοριακά προγράμματα. Αυτό είναι το τρωτό σημείο του FC. Ε, Δεν μπορεί η ΕΤΕ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, να χρηματοδοτήσει προς το πάνω διασυνοριακά προγράμματα και είπα ότι θα μπορέσουμε τα τις πολυεθνικές προτάσεις πλέον να τις προσεγγίσουμε, να τις χρηματοδοτήσουμε. Αυτή είναι νέα, εντελώς νέα προσέγγιση. Δεν υπήρχε νωρίτερα. Ε, και μπορούμε να ακούσουμε διάφορες απόψεις υπέρ, κατά, όμως το, το γεγονό είναι ότι όλοι ε, καταβάλουμε σκληρές προσπάθειες για να βρούμε λύσεις, ε, διότι υπάρχουν δυνατότητες σε κάποιους διαδρόμους για να χρηματοδοτηθεί ολόκληρος ο διάδρομος. Το RTMS, παραδείγματος χαρή, και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε χρησιμοποιήσουμε αυτή την πλατφόρμα για ένα ολοκληρωμένο δίκτυο. Θα ήταν τέλειο αυτό. Όμω αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε διότι δεν υπάρχει πλαίσιο θεσμικό για να γίνει αυτό. Και όπω σα είπα ενδεχομένω στο Ρότερνταμ να ε, μοιραστούμε μαζί σα καλέ ειδήσει ε, σε αυτόν τον τομέα. Επίση. και τα, οι χώρε συνοχή μπορούν ε, να ακολουθήσουν και να μάθουν ταχύτερα. Όπω είπα και στην αρχή μου ομιλία, δεν Υπάρχει ε, εκπαίδευση για τη χρήση των μηχανισμών του ΕΦΣΥ προς το παρόν. Ε, δεν υπάρχουν τρέχουσες πρακτικές, όμως ε, ας μην το δεχτούμε αυτό ως δεδομένο, να ανταλλάξουμε, να το συζητήσουμε με τους υπουργούς. Ε, εξακολουθούμε με τους εμπλεκόμενους φορείς των ε, κρατών συνοχής ε, να το συζητούμε και έχουμε κάνει την περιοδία μας, τα έχουμε εξηγήσει όλα αυτά και έχουμε προχωρήσει και γι' αυτό τώρα θέλουμε πιο στοχευμένες ποιοτικέ υπηρεσίες για να επισπεύσουμε τη διαδικασία εκμάθησης και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων καθώς και καλά παραδείγματα που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν και άλλοι φορείς, για να τους ενθαρρύνουμε δηλαδή. Αυτά είναι. Αυτή τη στιγμή... έχουμε επί τώρα και ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να κινηθούμε ταχύτερα ε, σε σχέση με τα όσα έγιναν κατά το παρελθόν, διότι αυτό είναι πραγματική πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τώρα, το ΕΦΣΙ είναι ένα, μια πρώτη προσπάθεια ανταπόκρισης. Μας ενδιαφέρουν μηχανισμοί που θα, θα θεμελιώσουν το έργο τους στην προηγούμενη εμπειρία πρέπει εδώ να υπάρξει καινοτόμος μηχανισμός ή συνέχεια του μηχανισμού αυτού με καινοτομία το βλέπουμε αυτό σε σχέση ε, με τις ε, δοκιμές που γίνονται πειραματικά με ένα νέο φόρουμ όπου ε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδυάζονται για τις μεταφορές. Πρέπει όμως αυτό να γίνει. Αγαπητέ Ντομινίκα, βασίζομαι σε σένα και σε πολλούς άλλους συναδέλφους που ενδιαφέρονται σε τέτοιου είδους πρότυπα χρηματοοικονομικά και με ανοιχτό πνεύμα τοποθετούμε. Σας δίνω την υπόσχεση ότι θα δώσω μάχη για τις μεταφορές. Βοηθήστε μας να υπάρξουν καλά θεμέλια, καλά πρότυπα που θα ακολουθηθούν. Αν θέλετε να πορευτούμε ταχύτερα, πρέπει από κοινού να πορευτούμε να κινηθούμε ταχύτερα, όλοι μας. Λοιπόν, τούτων λεχθέντων διασυνοριακά προγράμματα, διασυνοριακές ε, τέτοιες προσπάθειες, συνοχή. Συμφωνώ απόλυτα, με κάποια απογοήτευση βέβαια, όσον αφορά τους πολλαπλασιαστές ε, σε σχέση με τα προγράμματα αυτά. Ελπίζαμε να έχουμε πολλαπλασιαστές σε δεκαπλάσιους ή δεκαπενταπλάσιους όμως έχουμε διπλάσιους ή τριπλάσιους πολλαπλασιαστές αυτή τη στιγμή από πλευράς μόχλευσης. Δεν ε, προσελκύσαμε τα αναγκαία πιο θετικά αποτελεσματικά προγράμματα σε σχέση με την ε, δυνατότητα υποστήριξης μέσω χρηματοδότησης και επιδοτήσεων. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι κίνητρα που θα δοθούν και θα υπάρξουν ώστε να ενημερωθούν το δυνατόν ε, περισσότεροι, το ευρύτερο κοινό να κινητοποιηθούν και να συμμετάσχουν άνθρωποι που ποτέ δεν συμμετείχαν κατά το παρελθόν. Άνθρωποι που ποτέ δεν είχαν εξετάσει τη δυνατότητα να εμπλακούν και να συμμετάσχουν στον τομέα των μεταφορών. Βασιζόμαστε πολύ σε αυτή τη συνδιάσκεψη σύνοδο στο Ρότενταμ όπου άμεσα θα έρθουμε σε επαφή με ιδιωτικού επενδυτέ, με ιδιώτε επενδυτέ, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε περισσότερο τι απουσιάζει, κάποια στοιχεία που απουσιάζουν στοιχεία, για παράδειγμα όσον αφορά την φερεγγιότητα, τη ρευστότητα, για το πώς θα αντιμετωπίζονται ε, το, το επιχειρήν, πώς θα αντιμετωπίζεται. Δυστυχώς δεν γίνεται αυτό εν μια νυχτή και είναι επώδυνο για κάποιον που έχει ε, πνεύμα το επιχειρήν να αναμένει και να βλέπει τον χρόνο να παρέρχεται και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε αυτές τις διαδικασίες κάπως τουλάχιστον διότι το θέμα πραγματικά είναι φλέγον και ε, πρέπει να προαρθεί. Έχω ένα λεπτό ακόμη στη διάθεσή μου για το δίκτυο των ε, μεταφορών, των οδικών μεταφορών τοποθετήθηκα για το καμποτά, καμποτάζ και πάλι μέσα στο πακέτο μέτρων θα παράσχουμε, θα δώσουμε την επεξήγηση των κανόνων και ρυθμιστικών διατάξεων του Καμποτάζ. Ζητήθηκε να γίνει αυτό ήδη. Δεν υπάρχει ανάγκη για ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, για νέο νομοθετικό έργο, αλλά θα δούμε πού θα κινηθούμε και πώς. Ε, Στόχος μας είναι να συντμηθεί ο κύκλος ε, εργασιών και να είμαστε πιο ε, αποτελεσματικοί ταχύτερα να μπορούμε να δράσουμε σε έναν πιο σύντομο κύκλο δράσεων. Είναι μεγάλη η πρόκληση να μπορέσουμε να υποπτεύσουμε σωστά αυτό το θέμα. Το καμποτάζ είναι ένα θέμα που θα παραμείνει στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων υπό εξέταση και υπό συζήτηση. Στόχος μας είναι να καταλήξουμε σε μια κοινή επεξήγηση κανόνων και κανονισμών ώστε να μην υπάρχει αυτή η ποικιλία, η μεγάλη αυτή ε, ας το πω έτσι διαφορά μεταξύ των ερμηνεών που δίνονται πράγμα το οποίο είναι αντιπαραγωγικό. Σε σχέση τώρα με τα διόδια, σε σχέση με νέες, ε, ε, νέους δρόμους, αυτοκινητοδρόμους, ε, θα πρέπει ο χρήστης ανάλογα με τη συχνότητα τη χρήσης ε, του δικτύου να πληρώνει ανάλογα. Θα υπάρξει η εκπόνηση, η ανάπτυξη εκείνων των μέσων και εργαλείων ώστε να εισαχθεί αντικειμενικό στοιχείο ε, διαμόρφωσης διοδίων. Ε, όταν θα καταστεί αυτό δυνατό και αναγκαίο, ο χρήστης θα πληρώνει ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης του οδικού δικτύου. Με βάση αυτή την αρχή θα πορευθούμε και θα διαμορφώσουμε αυτά τα πλαίσια διοδίων. I'm uh, με ιδιαίτερη ικανοποίηση έχω την πρόθεση να μπορέσω να απαντήσω γραπτά σε όσους δεν μπόρεσα να απαντήσω και όσοι έχετε κάποια θέματα να τα αποστείλετε και θα τοποθετηθούμε από αυτόν και για τους σιδηροδρόμους να μην υπάρχει κάποια ανησυχία πολλά πράγματα θα γίνουν και πολύ ενδιαφέροντα Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ και για την παρουσίαση, για τις απαντήσεις και την προσφορά και για τις παρεμβάσεις που ε, θα τοποθετηθείτε και για τον διάδρομο 11 υπαριθμών 11 θα το κάνω εγώ ο ίδιος να δω αν υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή όχι. Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα που εκκρεμούν. Ο κύριος Φαντεκάμπ ήθελε να γνωρίζει ότι σε σχέση με τις υποσχέσεις που δόθηκαν για την επισκόπηση του Working Program, του προγράμματος εργασίας, εξαιρετικά πορευθήκατε και ε, δεν χρειάζονται εδώ πρόσθετες ε, επιστολές ή παρεμβάσεις. Μπορείτε εσείς να μας υποβάλλετε αυτά τα στοιχεία και να υπάρξουν τα τελικά στοιχεία Έχουμε τα στοιχεία για την Αυστρία. Ο Αλεξάνδρ Φαντεβέν είναι 53,3%, 49,7% ο αντίπαλός του. 30.000 είναι η διαφορά, 30.000 ψήφοι Μπορούμε να συγχαρούμε θερμά τον ε, νικητή των εκλογών και ελπίζουμε ότι στην Ευρώπη θα εξελιχθούν, θα μετεξελιχθούν τα πράγματα μέσα σε ένα θετικότερο πλαίσιο. Και έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ευχαριστώ και πάλι την κυρία Επίτροπο. Συνεχίζουμε αμέσως με το επόμενο σημείο, το 5 της ημερήσιας διάταξης. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. <laughs>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 take a seat. We will continue. Αφήστε παρακαλώ, θα συνεχίσουμε. Es geht jetzt über die Verordnung. Τώρα έχουμε τον κανονισμό για την δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Η συγγήτρια είναι η κυρία Αρνοτίου, έχει τον λόγο, παρακαλώ. Κυρία Αρνοτίου, έχετε τον λόγο. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, je vais, je vais être bref parce que... Ευχαριστώ και θα είμαι σύντομη Λυπάμαι, λυπάμαι πραγματικά ε, για αυτά που έγιναν στις 12 Μαΐου για το, την ψηφοφορία για το σχέδιο. Ήταν σοου, θλιβερό αυτό που συνέβη εδώ πέρα. Ε, και τι να πω, δεν άκουγαν πολύ, δεν είχαν διαβάσει την έκθεση, γιατί ε, ή δεν άκουσα τίποτα ή με προσβάλλανε ε, ε, ρατσίστρια με είπαν νομίζω ότι έχουν αποκοπεί πολύ από την καθημερινή ζωή των πολιτών. Γιατί πολλοί αντιμετωπίζουν καθημερινά τα προβλήματα της μαζικής μετανάστευσης και επισύρει αυτό προβλήματα ως προς την ταυτότητα, τη θρησκεία, την ασφάλεια, την οικονομική μας ζωή. Θα είμαι σύντομη γιατί τώρα που σας τα λέω αυτά Είτε μιλάμε από ιδεολογική ε, σκοπιά, είτε ε, το οποίο είναι και χειρότερο, όπω διαπίστωσε στι 12 Μαου, ανήκουμε σε κάποια κοινότητα, ε, δημιουργούνται αυτά τα θλιβερά φαινόμενα και δεν θα πρέπει να εκπλησώμεθα που στη Γαλλία τουλάχιστον λέμε ότι το πρώτο κόμμα σε δύναμη είναι η αποχή. Ναι, είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, αλλά να μην μα εκπλήσει μετά η δυσαρέσκεια εναντίον των πολιτικών, διότι οι συμπολίτε μα νομίζουν ότι ζούμε μέσα σε μια φούσκα. Θα κλείσω ε, ε λέγω, ζητώντας επίσημα από όλους σας ε, να να ξαναδιαβάσετε τις τροπολογίες, να τις λάβετε υπόψη, διότι είναι κοινή μας ευθύνη ε, σε σχέση με τους συμπολίτε μας και επίγει, επίγει να είναι ισχυρό το μήνυμα που στέλνουμε στα θεσμικά όργανα της Ένωσης ε, και το τονίζω εδώ γιατί μπορεί να παρερμηνευτεί, διότι καταπολεμούμε το θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σίγουρα όχι την Ευρώπη σε καμία περίπτωση. Ε, έχω την εντύπωση ότι μέσα στην οδηγία για το το νέο Frontex, ε, ε, αυτά που προτείνονται είναι ε, αμεληταία σε σχέση με τα πελώρια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και με αυτά τα πελώρια προβλήματα των μαζικών μεταναστευτικών νομών δεν επαρκούν αυτά τα στοιχεία του κανονισμού. Θα πρέπει λοιπόν να ξεπεράσουμε τα μικροκομματικά μας και να ε, βρούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ούτως ώστε να ε, δώσουμε μια άξια συνέχεια στην ιστορία μας, να τονώσουμε τη συνεργασία μας και νομίζω ότι εξάλλου αυτό είναι κοινός μας στόχος να ε, εξυπηρετήσουμε τον, τους λαούς της Ευρώπης να είναι σταθερό και βιώσουμε το πλαίσιο που τους προσφέρουμε για τις επόμενες δεκαετίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε εσείς. Ja, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μια ερώτηση. Είχατε την εντύπωση ότι θα ήταν εδώ η συγητής της Λίμπε. Ε, κάκουσα την κυρία Γνωτή, αλλά εγώ είχατε την εντύπωση ότι είχαμε μία, εν πάση περιπτώσει, σχετικά καλή ανταλλαγή απόψεων. Θα μπορούσα να τοποθετηθώ επί των όσων είπε. Αλλά επαναλαμβάνω ε, την ερώτησή μου. Ο εισηγητή τη Λίμπε θα είναι εδώ σήμερα. Der Ο εισηγητή τη Λίμπε είναι σε άλλη συνεδρίαση και δεν μπορεί να παραστεί αυτή τη στιγμή. Όταν θα είναι δυνατό θα προσέλθει. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Αύριο όμως θα διεξαχθεί η ψηφοφορία Φυσικά όταν έχουμε ψηφοφορίες για θέματα τα οποία θα αποφασίσει και η ΛΥΜΠΕ, γι' αυτό εγγράψαμε την ψηφοφορία για αύριο το απόγευμα. Όταν όμως προσέλθει θα μπορέσει να τοποθετηθεί. Ναι. Άρα μιλούμε για τον κανονισμό με τον οποίο ασχολείται η ΛΥΜΠΕ και όχι για την ε, γνωμοδότηση, αν κατάλαβα καλά. Δηλαδή ποιο είναι το αντικείμενο συζητούμε για το θέμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλειας Ναυσιπλοείας που συζητείται και από τη ΛΥΜΠΕ. Μάλιστα. Ε, κοιτάξτε Πρόεδρε, εγώ υποστηρίζω, υποστηρίζω θερμά την πρόταση της ε, Επιτροπής. Και αυτό είναι ένα σημείο από το οποίο συμφωνώ με την κυρία Αγνότου. Έχουμε μια τεράστια πρόκληση μπροστά μας, ένα πρόβλημα, να διαχειριστούμε την κρίση αυτή. Αλλά αυτή η έκθεση που συνέταξε η κυρία Αγνοτιού δεν είναι η θέση της Επιτροπής. Αναμειγνύει διάφορα ζητήματα εθνικού και θρησκευτικού χαρακτήρα που εμείς ε, δεν, δεν θα έπρεπε να τα εκφράζουμε κατά αυτόν τον τρόπο δεν θέλουμε να τα εκφράσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Θεωρούμε ότι πρέπει να τοποθετηθεί η Επιτροπή σε σχέση με την ΕΜΣΑ. Ακόμα άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη Μεσόγειο. Θα πρέπει να ληφθεί η δράση το συντομότερο δυνατό, άμεσα, και όσο πιο γρήγορα μπορέσουμε εμείς να ολοκληρώσουμε αυτή τη δουλειά, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσει να υλοποιηθεί και η φύλαξη των συνόρων. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου λοιπόν, σε πρώτη φάση. Ευχαριστούμε. Εσείς ευχαριστώ για τη σοσιαλιστική ομάδα τίθεται ως εξή το θέμα. Έχουμε μια σαφέστατη στρατηγική σε σχέση με την αντιμετώπιση αυτού του θέματος από την ομάδα μας. Κάθε τροπολογία θα την απορρίψουμε. Στο τέλος τέλος θα υπερψηφίσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί να αποστασιοποιηθούμε από κάτι το οποίο δεν θα είναι αποδεκτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αεφώτα, παρακαλώ. Yes, thank you very much, Chairman. Um, I think just for clarification. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χάρη διευκρίνησης για τις, τα στοιχεία που ανέφερε η κυρία Η πρώτη έκθεση που αναφέρθηκε ήταν για την εκτοφυλακή και εγώ εξήγησα υπό την οπτική του Ηνωμένου Βασιλείου και όχι της ομάδας ότι οι ομάδες που δεν είναι μέλη του Σέγγεν δεν θα συμμετείχαν βεβαίως θα συνεργαστεί το Ηνωμένο Βασίλειο στενά με τη Frontex η εντολή μας εκεί ήταν όμως ε, σαφώς διαφορετική τώρα για αυτήν εδώ την έκθεση συζητούμε εδώ εξετάζομαι τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του οργανισμού και επ' αυτού έχουμε δυσκολίες και περιπλοκότητες. Σε σχέση με την τελευταία συνάντηση, ίσως να μην συμφωνώ με τις απόψεις που εκφράστηκαν σε εκείνη τη συνάντηση από άλλα μέλη της Επιτροπής, αλλά πρέπει να είμαστε ευγενείς, είμαστε στα πλαίσια μιας κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, πρέπει να ακούσουμε τις άλλες απόψεις. Το καταθέτω και αυτό. Τώρα σχετικά με τη διεύρυνση του πεδίου της ΕΜΣΑ. Έχουμε όπως έλεγα ακαθόδη περιπλοκότητες σχετικά με τις δράσεις που θα αναλαμβάνει η ακτοφυλακή αυτή και σε σχέση με την εντολή της συγκεκριμένη τη ΕΜΣΑ. Εγώ υπέβαλα κάποιες ε, τροπολογίε που δεν ήταν καθόλου μικροπολιτικές αλλά στην τροπολογία 13 έπρεπε να αναφερθεί στο άρθρο 1 στα πλαίσια της εντολής, γιατί ο καθένας το κάνει διαφορετικό, οι, οι, οι λέξεις αυτές. Όπως και στη 15 για το 1-2. Ή υπό την προϋπόθεση συμφωνίας των ενεχομένων κρατών μελών. Εκεί. Γιατί η υπο την προυποθεση συμφωνια γνωρίζει πολύ καλά. Δεν είναι αφελής. Γνωρίζει ότι υπάρχουν δυσκολίες και ότι θα εξαρτηθεί από τα κράτη-μέλη σε πολλά σημεία. Η εκτοφυλακή στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν ασχολείται με θέματα μετανάστευση, σε άλλε χώρε ασχολείται. Επομένω, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν τη δομή που θα ασχολείται, που θα αναλάβει το κάθε τμήμα. Με αυτήν λοιπόν την υποσημείωση από πλευρά μου αναγνωρίζω ότι βεβαίω υπάρχουν αποκλήσει απόψει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της δημοκρατίας, ότι δεν είναι μοναδική αλήθεια κάποιου. Εσείς παρακαλώ στη συνέχεια, σας κουν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα εκπλήξει την εισηγητρία ούτε κανένα μέλος αν επαναλάβουμε την τοποθέτηση που προασπίσαμε σε μια προηγούμενη συνέδριαση που ήταν το ότι δεν θα καταθέταμε καμιά τροπολογία. Και καθώς αυτό το σημείο είναι η εξέταση των τροπολογιών, προαναγγέλλω ότι θα καταψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες που κατατέθηκαν και θεωρούμε ότι σε αυτή τη συγκυρία πρέπει να προσπίσουμε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την πρότασή της ως έχει. Και θεωρούμε εμείς ότι από τις ευρωπαϊκές αξίες πρέπει να ενδυναμωθεί αυτή η ευρωπαϊκή υπηρεσία. Διότι αυτή τη στιγμή δεν έχει τα εργαλεία και τους μηχανισμούς και τα αναγκαία μέσα που απαιτούνται για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Αυτό θα γίνει λοιπόν ανταποκρινόμενοι σε σχέση με την προαναγγελία που είχαμε κάνει. Αυτή θα είναι η θέση μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η σκιώδης εισηγήτρια της ΓΟΕ δεν παρίσταται. Εσείς θα παρέμβετε. Κιστέλα παρακαλώ. Thank you very much, Chair. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι διάβασα την έκθεση Αρνότου και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρέπει να πω ότι η έκθεση της κυρίας Αρνότου δεν αντανακλά την βούληση, την προτίμηση ή τον, την πρόθεση του κοινοβουλίου, του Κοινοβουλίου. Ιδιαίτερα σημειώνουμε την απουσία των, των όρων αναζήτηση, έρευνα και δικαιώματα του ανθρώπου και νομίζω ότι αυτό δεν την χάνει της πλειοψηφίας ε, του Κοινοβουλίου ως έχει και στην ε, Ευρωπαϊκή ε, Υπηρεσία Ασφάλειας δεν είναι μόνο το θέμα αυτό, δεν είναι μια πρόσθετη αρμοδιότητα απλώς. Ζητά η κυρία Αρνοτού να φανταστούμε τη ζωή των άλλων ανθρώπων και αναφέρεται κάνοντας αυτό το πώς ε, επηρεάζει τα, ε, η μετανάστευση της, ε, τη ζωή των ανθρώπων. Πρέπει όμως να διαρωτηθούμε τι γίνεται με τους ίδιους τους μετανάστες. Και το δηλητήριο με το οποίο η χολή με την οποία ε, αντιμετωπίζονται αυτά τα θέματα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Διότι αυτοί οι άνθρωποι, η, η, η, κατάσταση ε, της ζωής αυτών των ανθρώπων και των κινδύνων τους ε, είναι πραγματικά ε, έκδηλη. Και σε σχέση με τις τροπολογίες για το νομικό κείμενο το οποίο προτείνεται, και σε σχέση με την, ε, ε, τις προτάσεις αυτές από κοινού με άλλες, ε, η έκθεση της κυρίας Αρνοτού είναι απόλυτα απαράδεκτη. Και σε σχέση με την Επιτροπή είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουμε στη σωστή απόφαση και θα καταψηφιστεί αυτή όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσουμε αύριο. Πρόεδρο, σε ευχαριστώ. Και τώρα ο εισηγητής της Επιτροπής Λίμπε προσήλθε σε εμά. Έχετε τον λόγο λοιπόν παρακαλώ κύριε εισηγητά σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, σε σχέση με την τελευταία σύσκεψη των σκιωδών, ε, που δυστυχώ δεν ήμουν, θα ήθελα να πω ότι έρχομαι εδώ σε εκπρόσωπο ε, τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για την ε, νέα πρόταση για την ε, ακτοφυλακή, Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή. Σε τρεις εκθέσεις διαφορετικών επιτροπών μπορέσαμε να καταλήξουμε σε μία παράγραφο για τον Οργανισμό Ελέγχου της Αλίας, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θαλάσσιας Ασφάλειας και για την Ευρωπαϊκή Εκτοφυλακή. Λάβαμε υπόψη την γνωμοδότηση λοιπόν της Επιτροπής Αλίας, όμως από την Επιτροπή Μεταφορών δεν λάβαμε γνωμοδότηση. Και γι' αυτό είναι μάλλον γενικόλογη διατύπωση και φυσικά είναι συμβαστικό χαρακτήρα. Θέλω επίσης να τονίσω πως ε, Κάποιοι συνάδελφοι στην ε, Επιτροπή Μεταφορών ε, ρωτούσαν ή ανησυχούσαν, να το πω έτσι, για ποιο λόγο διαγράφει ένα σημείο στο 1β για ε, συστήματα τηλε, τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών. Ε, αυτό οφείλεται στη χρήση διότι είχαμε διάφορα παραδείγματα, drones ε, ή διάφορα αεροσκάφη, διάφορα πλοία και αποφασίσαμε από τη διατύπωση να τα διαγράψουμε όλα αυτά ε, για να τα καλύψουμε όλα. Δεν θέλαμε να ξεχάσουμε κάτι, θέλαμε να είναι ανοιχτό ο κατάλογος, ούτως ώστε να έχουμε τη βέλτιστη δυνατή χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού που θα έχει στη διάθεση των νέος αυτός οργανισμός. Αυτά ουσιαστικά από πλευρά μου και σας ευχαριστώ που μου δώσατε την δυνατότητα να εκφράσω την άποψη ε, από πλευράς Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Πρόεδρος, και πάλι σας ευχαριστούμε που προσήλθατε. Η Μπάρμπαρα Φαλιέ τώρα από τη Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής, παρακαλώ. Ναι, δεν θα μακρηγορήσω. Ε, θα επαναλάβω για τρίτη φορά κάποια πράγματα, δυστυχώς, και απαντώ στην κυρία Φώστερ λέγοντας πως ε, δεν είναι το θέμα μας η τροποποίηση του πεδίου για τους ε, τρεις οργανισμούς διατηρείται αυτό. Ενισχύουμε τις ικανότητε που έχουν και τη συνεργασία του, διότι ξέρουμε ότι η εκτοφυλακή έχει πολλές διαφορετικές λειτουργίες και η διοίκηση και οργάνωση των κρατών μελών διαφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό και γι' αυτό ε, προτείνουμε αυτήν την διπηρεσιακή συνεργασία. Θα σταματήσω εδώ γιατί το έχω ξαναπεί. Είναι κατεπίγον το ζήτημα και ο στόχος είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας ε, των ε, οργανισμών. Σας ευχαριστώ και πάλι τώρα η Μαρία Κριστίνα Αρναωτή, η συγγήτριά μας, για να κλείσει η συζήτηση. Κοιτάξτε, Πρόεδρε, ακούστηκαν τα πάντα. Εγώ δεν ξέρω τι μπορώ να προσθέσω ανησυχώ ακόμα περισσότερο που άκουσα δύο ομάδες που λένε ότι επί της αρχής δεν θα συμμετάσχουν. Δηλαδή αρνούνται είτε να υποβάλουν τροπολογίες είτε να το συζητήσουν ως θέμα αρχής. Αυτό το θεωρώ φοβερά ανησυχητικό για τη δημοκρατία, εγώ προσωπικά. Πάντως διατηρώ μια ελπίδα ότι αύριο θα εμφανιστούμε σε καλύτερο πνεύμα για το συμφέρον όλων. Αυτό απλώς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Όλοι συμφωνούμε λοιπόν να ξανασκεφτούμε αυτά τα θέματα μέχρι αύριο, διότι η ψηφοφορία θα είναι αύριο 24η Μαΐου 16 και 30. Και ολοκληρώνεται εδώ η επίσημη συνεδρίασή μας. Συνεχίζουμε και κλεισμένων των θυρών με τους συντονιστές. Χαίρομαι όταν αύριο 9 ακριβώς θα ξανασυναντηθούμε. Ναι και εσείς κύριε Φαντεκάμπ, 9 η ώρα ακριβώς.